first topic is the agenda. Hallo, guten Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste. Jetzt weiß ich auch. Χαίρετε αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι προφανές το γιατί χρειάστηκε να αναλάβω εγώ σήμερα την Προεδρία. Είναι τόση πυκνή κίνηση, το κυκλοφοριακό πρόβλημα στις Βρυξέλλες, ε, μετά τις ε, διακοπές φαίνεται και στους δρόμους ασφαλώς Γερμανίας, ε, που εκτός από τον κύριο Μπούσο, ή που εδώ και χαιρετίζω, δεν μπορούσε να έρθει και κανένας άλλος συνάδελφος. Φαντάζομαι ότι θα έχουν κολλήσει κάποιο μποτιλιάρισμα. Σε ξεκινήσουμε όμως με τις ανακοινώσεις. Έχετε λάβει τις προσκλήσεις, έχετε την ημερήσια διάταξη στα χέρια σας, υπάρχουν αντιρρήσεις. Ουχή. Χαίρετε κυρία Ρούλα και καλησπέρα. Καλώ ήρθατε, η μερική λοιπόν. Πρακτικά συνεδριάσεων τα έχετε λάβει και αυτά. 24-25 Σεπτεμβρίου, 10-11 Οκτωβρίου. Εάν ως το τέλος της συνεδριάσεως δεν κατατεθούν αντιρρήσεις στα πρακτικά, θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί. Έχω κάποιες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις επίσης. Όσοι ήθιστε. Καταρχάς, σας ενημερώνω ότι όσοι ήθιστε ε, ε, μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου η παρούσα συνεδρίαση. Επίσης, ε, έχουμε ένα μια αλλαγή στο προγραμματισμό μας 13 Νοεμβρίου από τις 3 έως τις 6 το απόγευμα θα γίνει η συζήτηση, η ακρόαση καλύτερα με τον υποψήφιο ο οποίος μάλιστα ονομάζεται Dr. Tony Bock, ο οποίος πρόκειται να αντικαταστήσει τον Επίτροπο κύριο Ντάλη. Την ακρόαση οργανώνουμε από με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τη Γεωργική Επιτροπή. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς θα έχει περίπου 30% του χρόνου της συνεδριάσεως, της ακροάσεως στη διάθεσή της, προκειμένου να διατυπώσουν τα μέλη της τις ερωτήσεις τους. Επίσης, η Γραμματεία της Επιτροπής μας καλωσορίζει ένα νέο συνεργάτη, τον κύριο Μπέγκιτάτ από την Γερμανία. Καλώς ήρθατε. Την κυρία Μπέγκιτάτ. Έχετε, νομίζω, ήδη γνωριστεί με όλα τα μέλη της Επιτροφής. Και τώρα περνάω στην ημερήσια διάταξη με την έκθεση του κυρίου Πουσόη. Εκ των σκιωδών παρούσα είναι η κυρία Ρούλα η κυρία Κάινα. Πολύ ωραία κύριε Μπουσόη. Μπορείτε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε που κατάσταν τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ για την συμβολή τους στην επεξεργασία του κειμένου. Λόγω της λεγόμενης πράσινης εβδομάδα δεν είναι στη δυνατή οργάνωση με πρόβλεψη μια συνεδρίασης ε, συντον... σκιωδών εισηγητών ε, την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά μείναμε σε επαφή μέσω των ε, βοηθών μας, του προσωπικού μας και πιστεύω ότι εν τέλει θα καταλήξουμε σε ένα καλό κείμενο. Θα ήθελα να σχολιάσω εν συντομία στις τροπολογίες και αν μου επιτρέπετε συνέχεια να ακούσουμε και τους συντονιστές. Έχουμε λοιπόν ε, τροπολογίες που στόχο έχουν να τροποποιήσουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας όσον αφορά τις συμβατικές συμφωνίες. Τώρα συμπεριληφθούν λοιπόν οι συμβατικές συμφωνίες στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας όταν πρόκειται για το μόνο τρόπο για την εισαγωγή ενός φαρμάκου στο σύστημα υγείας ε, και της νομοποίησης, της τακτοποίησης των ε, θεμάτων των σχετικών με τον αδιούχο. Ε, Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει αντίρρηση. Για τα βίο ισοδύναμα επίσης η τροπολογία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Για τις τροπολογίε υπάρχουν, υπάρχουν για τις χρολογίες μάλλον έχουμε μία τροπολογία η οποία προτείνει σε 30 ημέρες την ημέρα για την ε, έγκριση των βιοεισοδυνάμων, ε, γιατί θεωρείται ότι ανάλογα και με τα συνθήκε που ισχύουν σε διάφορε χώρε μέλη, μπορεί 15 μέρε να είναι πολύ σύντομη προθεσμία. Γι' αυτό και εγώ υπογραμμίζοντα ότι πάντα πρέπει να προσαρμοζόμαστε στι πρακτικέ, στι πραγματικέ συνθήκε, συμφωνώ. Βεβαίω θα πρέπει πάντοτε να γίνεται η αξιολόγηση τη υγεία και ασφάλεια ε, σε περίπτωση που είναι γνωστά τα δεδομένα, μπορεί να είναι πιο σύντομη η προθεσμία. Το άρθρο 7 για την ενσωμάτωση του, ε, του φαρμάκου του ισοδυνάμου στο, στο σύστημα υγείας ε, είναι ικανοποιητική. Η εξασφάλιση της διαφάνειας και της έγκαιρης πρόσβασης σε φάρμακα για τον Ευρωπαίο ασθενή νομίζω είναι μια πολύ σημαντική αρχή. Το άρθρο της σιωπηρής αδειοδότης του άρθρου 3 δεν νομίζω ότι πρέπει να το ξανασυστήσουμε. Το ίδιο η υποχρέωση για αιτιολόγηση των αποφάσεων με βάση τους στόχους και τα επιβεβαιώσιμα ή επαληθεύσιμα κριτήρια. Ε, πρόκειται εδώ για τροπολογίε δηλαδή οι οποίε μπορεί να μα οδηγήσουν σε όπιστο δρόμηση περισσότερο και να αποστείλουν πολύ ασφαλμένο πολιτικό μήνυμα ιδιαίτερα ως προς το ζήτημα της διαφάνειας και της υποχρέωσης για τα κράτη-μέλη να σέβονται τις, οδηγί... τις ε, διατάξεις. Το κομμάτι που αφορά την προσωρινή αναφορά, επίσης δεν είμαι, σαφή, ε, δεν είμαι σίγουρος αν το έχω καταλάβει ως προς το, την το προσωρινό πάγωμα των τιμών. Δεν ξέρω αν αυτό αφορά την τιμή την ίδια αν είναι λοιπόν προσωρινή η ιδέα, εν το, η ιδέα είναι το προσωρινό πάγωμα της, αγο... της τιμής, ε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά θα παρακαλούσα την κυρία Πιτικά είναι την κυρία Μπεράκη να μου το εξηγήσουν. Για την 75, τροπολογία της κυρίας Πρέντεκαστ. Ε, θεωρώ ότι ξεπερνά τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τις υποχρεώσεις διαφάνεια με την υποχρέωση για ε, δημοσίευση δηλώσεων συμφέροντο ω προ τη λήψη αποφάσεων. Νομίζω ότι πρόκειται για σημαντικέ αποφάσει. Αποφάσει οι οποίε ενδέχεται να εμφανίσει τη σύγκρουση συμφερόντων και ω εκ τούτου θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα τη τροπολογία. Στο 82 νομίζω δεν είναι καλή ιδέα η διαγραφή ολόκληρου του άρθρου. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσω είναι υπερβολική και γι' αυτό μπορώ να δεχθώ την διαγραφή των οικονομικών ε, τομέων και σε πνεύμα συμβαστικό προτείνω να διαγραφεί και το κομμάτι σχετικό με τις ζημίες που προτείνει η κυρία Πρέντεγκαρστ και να εισαχθεί μια παραπομπή στο αρμόδιο σώμα εφόσον δεν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Άρθρο 13 και στοιχεία που έχουν ήδη ε, αξιολογηθεί από τις σχετικές αρχές. Υπάρχουν ε, ε, συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν να εντοπίσουν κάποιες ομοιότητες στα κείμενα. Εγώ έχω αντίστοιχο κείμενο στο 99, μόνο όμως για τα ορφανά φάρμακα, για τον προσδορισμό των ορφανών φαρμάκων. Θεωρώ ότι 99 είναι ευρύτερη λοιπόν τροπολογία και γι' αυτό παρακαλώ να την υποστηρίξετε και να υποστηρίξετε και, τον, ε, και την αλλαγή στην επικεφαλίδα ώστε να είναι πιο σύντομη. Άλλο ένα άρθρο με την είναι αυτό του με τον αριθμό 16 για την κοινοποίηση των σχεδίων μέτρων. Σημαντικό άρθρο, διότι δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαρκή ενημέρωση για τα μέτρα και τη δυνατότητα για εκκίνηση διαδικασία επί παραβάση, εφόσον χρειαστεί αυτό. Βέβαια, εδώ υπάρχουν αντιρρήσει και επιφυλάξει από κάποιου συναδέλφου που θεωρούν ότι είναι επικίνδυνη η επιβάρυνση με πολλέ διαδικασίε των κρατών μελών. Γι' αυτό θα πρότεινα εγώ μια πιο ήπια διατύπωση και θα προτείνω εγώ στο σχέδιο γνωμοδότηση μια μικρή τροποποίηση ότι δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από την υιοθέτηση των μέτρων. Εν τέλει δε, κάποιες τροπολογίες που αφορούν τη διαφάνεια στις τιμές. Η οδηγία ασχολείται με την διαφάνεια της λήψεως αποφάσεων σχετικά με τις τιμές αυτή καθεαυτή και όχι με τις ίδιες τις τιμές. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε ανταγωνιστικότητα και η διαφάνεια των τιμών ε, βεβαίω είναι πολύ καλή ιδέα, αλλά μπορεί να έχει κάποιε απρόβλεπτε επιπτώσει προ την ε, βιωσιμότητα όλου του συστήματο και με λίγα λόγια θα το εξηγήσω πριν ε, ολοκληρώσω. Η διαφάνεια των τιμών μπορεί να οδηγήσει σε σύγκληση των τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει και τη αρχή τη ενιαία αγορά. Αλλά δυστυχώ δεν υπάρχει ακόμη στα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα είναι η αγορά και θέλω αυτόν τον λόγο ότι τα συστήματα υγεία είναι διαφορετικά, τα, εισοδήματα, τα επίπεδα, τα οικονομικά των κρατών μελών είναι πολύ διαφορετικά και ω εκ τούτου είναι πολύ διαφορετικές τιμέ που καταβάλουν οι ε, ασθενεί από την ε, μία χώρα στην άλλη. Και έτσι υπάρχουν ε, ασθενεί στι χω... χώρε για του οποίου είναι χαμηλότερε τιμέ των φαρμάκων και σε άλλες χώρες πιο πλούσιες είναι πιο ε, υψηλές τιμές των φαρμάκων. Αυτό μπορεί να επηρεάσει λοιπόν εάν οδηγηθούμε σε σύγκληση προς τα άνω μπορούμε να οδηγηθούμε σε πολύ, σε πολύ ακριβότερες τιμές φαρμάκων εις βάρος των φτωχότερων ε, κρατών. Αν ε, η τάση όμως είναι αντίστροφη τότε θα μειωθεί το περιθώριο κέρδους και ως εκ τούτου η πρόσβαση στα φάρμακα για όλους μας. Ο μόνος που μπορεί να κερδίσει από την διαφάνεια στις τιμές, από την υποχρεωτική διαφάνεια στις τιμές, είναι όποιος αναπτύσσει παράλληλο εμπόριο στα φάρμακα, που δυστυχώς γνωρίζουμε ότι υπάρχει, κυρίως από τις χώρες με χαμηλές τιμές προς τις χώρες με υψηλότερες τιμές. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να μην επιμείνουν οι συνάδελφοι με τις τροπολογίες για τη διαφάνεια στο σχηματισμό των τιμών. Ε, επίσης καλώ τα κράτη-μέλη με μια δική μου τροπολογία να ε, επιλέγουν στον, για το σχηματισμό της, για τη λήψη απόφαση και με την τιμή να επιλέγουν ε, ως μέτρο σύγκρισης κράτη-μέλη με αντίστοιχο οικονομικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Και στη διάθεσή σας αν χρειάζεται κάτι. Κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βουσόη. Δύο σκιώδεις είναι παρόντες εδώ. Ας ξεκινήσουμε με την κυρία Πίτι Κάιναν και μετά η κυρία Ρούλα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Μπουσόη για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Αν και έγινε ε, λίγο έτσι με κάποια ψηλοεμπόδια λόγω της Πράσινης Εβδομάδας και πιο πολλοί συνεργάτες μας ήταν αυτοί που δούλεψαν, αλλά ήταν πολύ επικοδομητική η συνεργασία μας παρόλα αυτά. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δική μας γνωμοδότηση και τη δική μου γνωμοδότηση, δεν βλέπω να υπάρχουν ε, μεγάλες ε, διαφορές ε, μεταξύ των Ευρωβουλευτών και μεταξύ των κρατών μελών. Εντάξει, υπάρχουν διαφορετικά πολιτικά κόμματα, αλλά νομίζω ότι παρόλα αυτά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να γεφυρώσουμε τις θέσεις ε, του Συμβουλίου που ήταν ε, άκρος αρνητικό για την όλη πρωτοβουλία συνολικά με τις πληροφορίες που έχουμε όλοι δηλαδή ότι ακόμη και για το πάγωμα της δικασίας αναθεώρησης ε, είναι μια τακτική και εμείς προσπαθούμε με το δικό μας τρόπο, με πολύ συνετό τρόπο νομίζω, να δημιουργήσουμε κάποιες εξελίξεις τελικά και να μετακινηθεί και το Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, πράγματι νομίζω ότι πολύ καλά προβλέπετε εσείς ε, νέες ε, προθεσμίες. 60-120 μέρες και για τα νέα φάρμακα 180 μέρες και για τα κοινόχρησης ονομασία στα γενώσιμα. Εκεί έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα με αρκετά κράτη-μέλη. Οπότε εκεί εγώ θα πρότεινα να υιοθετήσουμε την προθεσμία των 30 ημερών και θα ήθελα να ακούσω και τα σχόλιά σας. Συμφωνώ επίσης με την ανάλυση σας για το άρθρο 16. Διότι και εγώ σκεπτόμουν ότι αυτό συνεπάγεται μεγάλο γραφειοκρατικό βάρο για τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να σταθμίσουμε τα υπέρ και τα κατά σε ό,τι αφορά την αύξηση της γραφειοκρατίας για τις κοινοποίησεις από τα κράτη-μέλη. Καλό θα ήταν να αξιοποιείται καλύτερα ο χρόνος. Πάντω ε, θα το μελετήσω, θα μπορούσαμε να το αφήσουμε ανοιχτό και να δούμε τι είδου συμβιβασμό μπορούμε να βρούμε και με τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο. για τη μη παρέμβαση, για τα θέματα ασφάλειας των ασθενών κτλ. Υπάρχουν κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τη διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ίσως θα ήταν καλύτερα να λέμε κριτήρια και όχι στοιχεία, κριτήρια όχι elements, αλλά δεν ξέρω, μπορούμε να εξετάσουμε και ίσως και κάποια αναλλακτική διατύπωση, γιατί ο στόχος μας είναι να είναι εγγυημένη η πρόσβαση σε ερευνητικό υλικό από την διαδικασία της χορήγησης άδεια κυκλοφορία. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσει, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό το σκέλος. Δύο από τα μείζωνα ζητήματα και εκεί παρατηρώ και τις ε, μεγαλύτερες διαφορές στις δύο γνωμοδοτήσεις, είναι αυτή η δική σας ε, πρόταση στο άρθρο 5 για προσωρινό πάγωμα τιμών. Και έχουμε και ε, μια προσπάθεια να μειωθεί το γραφειοκρατικό βάρος για τα κράτη-μέλη. Διάφορες διαδικασίες, ανακοίνωσης Όταν μιλάμε για μεταφορές, price transfers, καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν αναρμονίζουμε όμως, δεν ε, προσπαθούμε να κάνουμε εναρμόνιση στις τιμές, ε, στην τιμολόγηση, άρα πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια κατά την απόψη μου στις τιμές. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και σε επίπεδο κρατών μελών λοιπόν με την τιμολόγηση των φαρμάκων, γιατί είναι και προ όφελο των ασθενών. Μια βάση δεδομένων για τις τιμές των φαρμάκων είναι μια ε, πρόταση αξιοσημείωτη που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πολύ σύντομα εγώ, κυρία Ρούλα. Υποστηρίζω εν γέννη τον εισηγητή και τα όσα μας παρουσίασε. Μια ερώτηση μόνο, ίσως όμως να μπορούμε να το, λύσουμε διμερώς εκ των υστέρων. Για την 74 της κυρίας Βερνιό, τι γνώμη έχει ο εισηγητής, γιατί εμένα με δυσκολεύει η πρόταση να πρέπει τα κράτη-μέλη να δημοσιεύουν κατάλληλα ή επαρκή ποσά πιστώσεων και να εξηγούν ε, εάν πρόκειται για φαρμακευτικά προϊόντα στο χώρο της ασφάλισης ή όχι. Νομίζω ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρωτάει τα κράτη-μέλη στις πιστώσεις αυτές ποιο κομμάτι πάει στην, ε, στην κοινωνική ασφάλιση. Ε, λέτε ότι το καταψηφίσετε. Πολύ καλά. Είσαστε κατά, κατά της διαγραφής. Είσαστε κατά της τροπολογίας. Πολύ καλά λοιπόν, θα συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βάιλερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τώρα το εξή δίλημα ότι μας περισσεύει λίγος χρόνος. Κύριε Μπουζόη, θέλετε, μια και έχουμε χρόνο πριν να λάβετε το λόγο εσείς για τελικά σχόλια, να ακούσουμε την Επιτροπή, αν υπάρχει κάποιος εδώ. Θέλει η Επιτροπή. Μια και έχουμε χρόνο, ο κύριος Σουάπ δεν έχει έρθει ακόμη. Θέλετε τώρα να μιλήσετε, αργότερα. Όχι, καλώς. Κύριε Μπουζόη. Αν θέλετε να δώσετε κάποιες απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα μου πάρει πάνω από δύο λεπτά. Ο κύριος ε, Σβάμπ, ως Γερμανός είμαι βέβαιο ότι θα είναι εδώ, ε, βέβαιος ότι θα είναι ακριβώς την ώρα του στις 3.30 εδώ. Λοιπόν, καταλαβαίνω την κυρία Πιτικάινεν και θέλω να την ευχαριστήσω για την επικοδομητική της προσέγγιση και γιατί κατανοεί τη θέση μας ε, σε ό,τι αφορά τα ε, γεννόσιμα φάρμακα και είναι ένα ζήτημα το οποίο θέτουν στο Συμβούλιο ορισμένα κράτη-μέλη, άρα 30 ημέρες δεν είναι και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι σημαντικό να είναι σαφείς οι προθεσμίες αλλά και εφικτές, γιατί θέλουμε να υλοποιηθεί πραγματικά η οδηγία αυτή. Σε ό,τι αφορά την διαφάνεια στις τιμές, το καταλαβαίνω και αυτό και φαντάζομαι ότι και οι συνάδελφοι καταλαβαίνουν και τη δική μου θέση. Προέρχομαι από ένα νέο κράτος μέλος όπου οι τιμές εκεί ίσως είναι χαμηλότερες από τις άλλα κράτη-μέλη. Πάντως καταλαβαίνω ότι η απόπειρα αυτή, δηλαδή να προχωρήσουμε προς την ίδια κατεύθυνση όλοι, θα μπορούσε να έχει και κάποιες ε, ανεπιθύμητες ε, ενέργειες, δυσάρεστες επιπτώσεις. Τώρα, για την κυρία Ρούλε, δεν είμαι και τόσο υπέρ της τροπολογίας της κυρίας Βερνιό. Αλλά θα προσπαθήσω να το συζητήσουμε διμερώς με την κυρία Βερνιό και να δούμε ακριβώς για ποιο λόγο έχει κάνει αυτή την πρόταση. Δυστυχώς χθες δεν είχαμε και πολλές συμβαστικέ προτάσεις. Όποτε στο παρελθόν διατέλεσα εισηγητής, ξέρετε ότι πάντοτε προσπάθησα να εξεύρω στον περισσότερους συμβιβασμούς το ζήτημα είναι πολύ λεπτό και φυσικά ε, συντάσσουμε γνωμοδότηση όλοι μας για την Επιτροπή ΕΜΒΗ, την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Επειδή όμως υπάρχουν πολλές τροπολογίες, ένας μεγάλος αριθμός τροπολογιών, δεν θα είναι και τόσο εύκολο να ικανοποιηθούν άπαντες. Θα προσπαθήσουμε όμως. Γιατί το σημαντικό είναι να προχωρήσουμε με την οδηγία αυτή. Και μετά την έγκριση της οδηγίας, δεν θα έχουμε σημερινές ε, καταστάσεις, δηλαδή να έχουμε κάποιες καταστάσεις, καταλόγους ε, ε, φαρμάκων ε, που, για τα οποία υπάρχει επιστροφή εξόδων και να μην έχουμε επικαιροποίηση του καταλόγου για τέσσερα χρόνια, για παράδειγμα, γιατί ισχύει αυτό για κάποια κράτη. Ευχαριστώ πολύ. 10 ώρα αύριο το πρωί λίγη προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών. Ο κύριο Σβάπ, όπω ε, ακούσατε κύριε Σβάπ, ε, ε, σώσατε τη γερμανική φήμη γιατί είσαστε συνεπέστατο Γιατί έλεγε πριν ο κύριος Μπουσόη ότι θα έρθετε ακριβώς στις 3.30 και το πράξατε. Μπράβο σας. Μπορείτε λοιπόν να ξεκινήσετε τώρα με τη δική σας έκθεση. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι οι γερμανικές ορογραμμές ευθύνονται και έτσι κατάφερα να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Συνάδελφοι, ένα πολύ σύντομο σχόλιο ενίδη για την ετήσια έκθεση περί ανταγωνισμού. Και τη γνωμοδότηση της δικής μας Επιτροπής για την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Θα πρέπει εδώ να επικεντρωθούμε στις ε, βασικές αρμοδιότητές μας για συγκεκριμένα ζητήματα. Γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ και στα τέσσερα ζητήματα που είχαμε τονίσει πέρσι και να δούμε ότι φέτος τα τέσσερις προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από τροπολογίες όσον αφορά την διάρκεια και την ακρίβεια της εκθέσεως η 40η επέτειος της εκθέσεως για την εσωτερική αγορά και της επιχείρησης που δραστηριοποιούνται σε αυτή βεβαίω, είναι πάρα πολύ σημαντική και την χαιρετίζουμε. Στην Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς λοιπόν θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τέσσερα κυρίως θέματα. Τέσσερι τομεί που ενδιαφέρουν πιστεύω και του συναδέλφου για την πολιτική ανταγωνισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τους καρόνες του ανταγωνισμού, έτσι ώστε και στο μέλλον ο καταναλωτής στην εσωτερική αγορά να έχει τη θέση του και ένα πλαίσιο ε, κανονιστικό. Ένα τομέα λοιπόν που ταχύτατα αναπτύσσεται είναι αυτός του e-payment, των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η αγορά αυτή, ο τομέας αυτός, για άλλη μια φορά, έχει ε, χαρακτηριστικά κατακαιρματισμού μέσα από τις τράπεζες, μέσα από τα κράτη-μέλη. Και αν μπορέσουμε, όπως ε, άλλωστε είχαμε αποφασίσει και στην έκθεση του συναδέλφου Αρίας, να εξετάσουμε με την ε, ηλεκτρονική αγορά, θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση αυτού του του σημαντικού κατακαιρματισμού της ε, αγοράς, του τομέα των ηλεκτρονικών αγορών, πληρωμών καλύτερα και άρα θα έχουμε καλύτερες συνθήκες. Δεύτερο σημείο, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, έχει να κάνει με τις μεταφορές εξπρές τις λεγόμενες, αερομεταφορές κυρίως, όπου πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει ε, μια ενδεχόμενη συγχώνευση στον τομέα αυτών. Θα έχετε ασφαλώς διαβάσει και από τον τύπο ότι υπάρχουν προσπάθειες από πλευράς της Αμερικανικής εταιρείας UPS να εξαγοράσει την TNT, Ολλάνδο-Βελγική ε, εταιρεία αερομεταφορών, ταχυμεταφορών. Δεν μιλούμε για συγχώνευση μεγάλων ε, ε, εταιριών στην, ε, στις ταχυμεταφορές. Ωστόσο, εμείς έχουμε διατυπώσει επιφυλάξεις με την έννοια ότι μια σειρά αγορών μπορεί να βρεθούν πλαγίως ή εμέσως εξαρτωμένων αγορών μπορεί να βρεθούν σε εξάρτηση από μονοπωλιακή σχέση. Γι' αυτό πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει αυτή τη συγχώνευση και εις βάθος. Τα, επίσης, εξετάζουμε και με την έκθεση του κύριου Έγγελ για την εσωτερική αγορά την ε, περίπτωση κατά την οποία ε, στη διεθνή αγορά, ειδικότερα σχέση με τις αμερικανικές επιχειρήσεις, ότι δεν έχουμε αντίστοιχη δυνατότητα πρόσβασης για τις δικές μας επιχειρήσεις. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να εξασφαλίσουμε συνθήκες ισότιμες για την πρόσβαση των επιχειρήσεών μας στην Αμερικανική αγορά. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη είναι μια σημαντική αγορά για τους Αμερικανούς, αλλά δεν διστάζουν παρόλα αυτά να ε, εγείρουν σημαντικά εμπόδια στην ε, παρουσία ιδιαίτερα στον τομέα των αερομεταφορών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ε, στι ΗΠΑ. Το είδαμε συγκεκριμένα με την Deutsche Post, η οποία τελικά αναγκάστηκε να παρετηθεί από μια τέτοια προσπάθεια. Το Evergreen τώρα είναι ο ιδιωτικό τομέα, πρόκειται για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργεια. Ο Επίτροπο κατέθεσε το τρίτο πακέτο, το οποίο υποστήριξε το Κοινοβούλιο πριν από μερικού μήνε μόλι, και εδώ έχουμε να κάνουμε και με την ε, ε, οδηγία για τι παραχωρήσεις Εάν λοιπόν αυτό το πακέτο μέτρων ε, υιοθετηθεί, θα, έχουμε, θα εξασφαλίσουμε στην αγορά ενέργειας μια ανοιχτή αγορά, μια ελεύθερη αγορά, αλλά αυτή θα πρέπει βεβαίως να εξασφαλίσει επαρκείς δυνατότητες ε, επιλογής για τον καταναλωτή πάνω απ' όλα. Εάν ανοίξει αυτή η αγορά ενέργειας, ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλιστούν και ισότιμες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ενεργείας, ε, αυτό ήταν ο τρίτο τομέα. Και ο τέταρτο και τελευταίο σημείο τη εκθέσεω έχει να κάνει με την αυτοκινητοβιομηχανία, με την αγορά μάλλον του αυτοκινήτου και την ε, πώληση ε, νέων οχημάτων από τον έμπορο πέραν του μέχρι τώρα ισχύοντος συστήματος του αποκλειστικού αντιπροσώπου, ενός συστήματος το οποίο είναι πολύ ε, ακριβό το οποίο σε συνθήκε κρίση και ιδιαίτερα στο χώρο του αυτοκινήτου πρέπει να μετατραπεί πλέον, πρέπει να ε, εξελιχθεί έτσι ώστε να μειωθεί και το κόστος για τον έμπορο. Έτσι πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιμείνει ως προς την ε, διατύπωση βασικών αρχών και σε περίπτωση κατακόρυφων συμφωνιών μεταξύ παραγωγού και εμπόρου στο χώρο των οχημάτων με όρους διαφάνειας τόσο για τις εμπορικές όσο και για τις συμβατικές σχέσεις. Από τη μία παραγωγός, από την άλλη έμπορος. Κυρία Πρόεδρε, αυτά τα τέσσερα σημεία η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων έχει ε, ήδη ξεκινήσει την εξετάσταση του θέματος. Δεν ξέρω τι πίεση χρόνου έχουμε από τη δική μας την ε, πλευρά για τη γνωμοδότηση. Θα μου πείτε εσείς. Ευχαριστώ κύριε δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση ουσιαστικά γιατί οι επισήμω οριστέντε ω και ο δεν είναι παρόντε. Δεν ξέρω αν κάποιο άλλο εκπρόσωπο πολιτική ομάδα θέλει να λάβει το λόγο. Ο κύριο Μπουσόη, εκ μέρου των φιλελευθέρων, ενδεχομένω θέλει να ε, ε, αντικαταστήσει τον κύριο Χατζημαρκάκη. Όχι. Οι πράσινοι νομίζω δεν έχουν ορίσει σκιώδη, ούτε εσείς. Η ECR δεν είναι παρούσα, η ΓΚΟΕ, η ΑΕΦΤ δεν είναι Για τους σοσιαλιστές δημοκράτες έχω γνωμοδότηση του κυρίου Κοφεράτη. Λάβει, δεν θα σας την αναγνώσω, νομίζω ότι δεν έχουμε τέτοιο περιθώριο, αλλά θα την διαβιβάσω με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους λοιπού σκιώδει, έτσι ώστε να γνωρίζετε ποια είναι η θέση των σοσιαλιστών δημοκρατών στην ε, γνωμοδότηση. Αλλά έχω και εγώ μία πρόταση, μια ερώτηση μάλλον, για το πρώτο σημείο, για τι ηλεκτρονικέ πληρωμές. Σω θα μπορούσατε να ε, μου δώσετε κάποιε λεπτομέρειε περαιτέρω, γιατί αν κατάλαβα καλά, ε, οι ηλεκτρονικές πληρωμές καρκινοβατούν και επειδή ο έμπορος εν γέννη επιβάλλει σημαντικό, ε, αντιμετωπίζει σημαντικό κόστος για την εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι ασφαλείς αυτές οι ηλεκτρονικές πληρωμές. Και αν δούμε τα άρθρα σε όλες τις, ε, ηλεκτρονικές, σε όλες τις σοβαρές εφημερίδες ε, που καταγγέλουν κινδύνους ε, να σπάσει κάποιος τον κωδικό πολύ εύκολα εν τέλει, νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη ασφάλεια Άρα, ασφαλώς στο μέλλον θα, μπορούμε να, θα, θα, θα δούμε κάποια στιγμή την ηλεκτρονική πληρωμή μέσω του κινητού τηλεφώνου, αλλά μέχρι τότε πρέπει είτε με μια ηλεκτρονική κάρτα ή με κάποιο άλλο σύστημα να εξασφαλιστεί ο όρος της ασφάλειας των συναλλαγών. Η κυρία Ρούιλε ζητάει το λόγο. Ναι, αν μου επιτρέπετε μια σύντομη παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σφάπ που συμπεριέλαβε και το θέμα των ε, αυτοκινήτων, των οχημάτων και την ε, ισορροπία δυνάμεων μεταξύ παραγωγού και εμπόρου, ένα ζήτημα το οποίο διαρκώς μας ε, προξενεί δυσκολίες στην εσωτερική αγορά. Υπάρχουν ζητήματα βεβαίως τα οποία δεν προχωρούν όπως θα θέλαμε και που οδηγούν σε στρέβλωση ανταγωνισμού μέσα στην εσωτερική αγορά, εις βάρος των πιο αδύναμων και ιδιαίτερα ε, σημαντική επιβάρυνση οικονομική στον χώρο της επισκευής των αυτοκινήτων. Ναι, και μία σύντομη συμπλήρωση. Ξέρω ότι προέρχεστε από κρατήδιο με μεγάλη παραγωγή αυτοκινήτου. Ο έμπορος πολύ συχνά δεν είναι καν ενήμερος των συνθήκων που ισχύουν στην εσωτερική αγορά. Ξέρετε ότι πολλές φορές μου λένε «Άμα αν πάτε με το αυτοκίνητο από εδώ εκεί ε, θα χάσετε τις εγγύσει σας». Ε, χωρίς ε, να είναι ενήμερος λοιπόν ο παραγωγός, ο ίδιος ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Καλό θα είναι μη τι άλλο να ενημερώνονται. Και πάντως το κοινοβούλιο είναι σε αυτόν τον αγώνα μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανείς άλλος. Όχι. Είναι όλοι ικανοποιημένοι με τις προτάσεις του κύριου Σφάπ για τις τροπολογίες. 27 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι έχει οριστεί η προθεσμία. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κύριε Σφάπ. 17 Δεκεμβρίου σύστομα τις τροπολογίες. Οχ. Και 18 ψηφίζουμε. Το που είπα ήταν γιατί δεν ξέρω, αυτές τις δύο μέρες μόλις πριν από τις ε, διακοπές των Χριστουγέννων θα έχουμε αρκετή προσέλευση. Η περισσότερη από ό,τι σήμερα, εν περιπτώσει. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα σημαντικών οδηγιών ασφαλώς, ασφαλώς θα υπάρξει επαρκής προσέλευση και φαντάζομαι ότι οι συντονιστές θα μεριμνήσουν αναλόγως. Γιατί βέβαια χωρίς σημαντική ε, πλειοψηφία από την Επιτροπή δεν είναι καλό να ψηφίζουμε ε, οδηγίες τόσο μεγάλου εισεμβέλειας και σημασίας. Άρα. Α, κύριε Σφάπ, ναι. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία αντίρρηση ως προς το θέμα των ηλεκτρονικών πληρωμών. Για να έχει ο καταναλωτής αυτήν ασφάλεια των συναλλαγών πρέπει να έχει τη δυνατότητα της ε, του να ξανασκεφτεί την πληρώμη. Πρέπει να ξέρουμε ωστόσο ότι υπάρχουν πολλοί καταναλωτές συγκριτικά που χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό με ολιγοπολιακή σχέση ως προς τις δομές εκείνες προσφέρουν ασφαλείς πληρωμές. είναι ε, εδώ συστήματα διαφορετικά από αυτά που έχουμε σε σχέση με τις ε, τράπεζες, επί παραδείγματι, ή τους παραδοσιακούς ε, παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Το κόστος μερικές φορές είναι αρκετά υψηλό και τα συστήματα ρύθμισης διαφορών μερικές φορές είναι πολύ δαπανηρά και δύσκολο να λειτουργήσουν σε ορισμένα κράτη-μέλη, ανάλογα με το κράτος μέλος. Άρα λοιπόν πρέπει με το νέο σύστημα να έχουμε μια ικανοποιητική προστασία και προσφορά υπηρεσίας για τον καταναλωτή, ώστε να μην διστάσει να προχωρήσει στην ηλεκτρονική πληρωμή. Για την κυρία Ρούιλε. Και τον χώρο του αυτοκινήτου συμφωνώ και πιστεύω ότι θα πρέπει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ελεύθερης συμβάσεως, περί συμβατικής ελευθερίας μεταξύ εμπόρων και ε, κατασκευαστών αυτοκινήτων θα πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή γιατί βέβαια ο χώρος του αυτοκινήτου έχει μια πολύ διαφορετική δομή από ό,τι άλλοι, άλλοι ε, εμπορική. και το ζήτημα το σχετικό με τις επισκευές των οχημάτων θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ό,τι φαίνεται βλέπει τα κύρια προβλήματα στο χώρο των νέων, ε, των νέων αυτοκινήτων περισσότερο. Ευχαριστώ. Gut, danke Herr Schwab. Sie sehen die Verwaltung. Ευχαριστώ πολύ κύριε Schwab. Για τις τέσσερις έχει προβλεφθεί η επόμενη έκθεση. Φαίνεται ότι η διοίκηση εδώ, οι υπηρεσίε της Επιτροπής μας, ότι περιμένανε περισσότερες διαφωνίες ως προς την έκθεσή σας. Φαντάζομαι ότι θα έρθει ο κύριος Ζιβά. Άρα μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για καφέ. Δέκα λεπτάκια. you. Liebe Kolleginnen und Kollegen, αγαπητοί συνάδελφοι, Ich eröffne die unterbrochene Sitzung erneut. Μπορούμε να συνεχίσουμε την συνεδρίαση που είχαμε διακόψει πριν από λίγο. Οι εισηγητέ και μέγα τμήμα των σκιωδών έχουν επιτέλους φτάσει. Και έτσι περνώ στο σημείο 6 της εκθέσεως, την ε, έκθεση, συγγνώμη, για ε, τις συμβάσεις παραχώρησης με τον κύριο Ζουβέν. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω την τιμή λοιπόν να ξεκινήσω εγώ με τη συζήτηση επί των τροπολογιών για το σχέδιο έκθεσης ε, αυτής, ό,τι αφορά δηλαδή τις ε, συμβάσεις παραχώρησης, πάνω από 780 ήταν τροπολογίες ε, και είχαμε για άλλες 236 στο σχέδιο έκθεσης. Θα σας κάνω λοιπόν κάποιες συνολικές παρατηρήσεις. Δεν μπορώ να καλύψω κάθε μία ξεχωριστά όπως καταλαβαίνετε και μετά θα ακούσω και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η δουλειά αυτή είναι καρπός ε, πολλών ε, εβδομάδων ε, συλλογικής δουλειάς και με τους σκιώδεις συζητητές και με άλλους συναδέλφους. Καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο από κοινού και οι θέσεις μας ε, σιγά σιγά μετακινήθηκαν πιο κοντά, έχουμε προσεγγίσει. Δηλαδή πριν από ένα χρόνο ήταν πολύ πιο απομακρυσμένες οι απόψεις μας και τώρα έχουμε κάνει πολύ δρόμο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ε, τροπολογίες για το σχέδιο έκθεσης, ήδη ευρύνουν τις προτάσεις, διευρύνουν το πεδίο τους και νομίζω ότι τελικά στηρίζεται η κοινή μας προσέγγιση, δηλαδή για την αναθεώρηση επί της ουσίας του αρχικού κειμένου της ε, Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τέσσερις, έχουν κατατεθεί τέσσερις τροπολογίες για απόρριψη του κειμένου. Οι τροπολογίες αυτές για απόρριψη υπογράφονται από συναδέλφους διαφόρων πολιτικών ομάδων οι οποίοι θεωρούν συχνά ότι μια νομοθετική πρωτοβουλία για τις συμβάσεις παραχώρησης δεν είναι αναγκαία ή περιπλέκει αχρίαστα, συχνά ε, τίθεται αυτό το, ως επιχείρημα, περιπλέκει λοιπόν τις νομικές δομές που υπάρχουν σε κάποια φυσικό όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να υποστηρίξω τις τροπολογίες αυτές και ένα πράγμα μόνο θα επισημάνω για μια ακόμη φορά. Το σχέδιο έκθεσης που σας παρουσιάζω και προτάσεις που διατυπώνω τροποποιούν άρδιν, άρδιν την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προτάσεις αυτές νομίζω είχαν απλουστευτεί και σήμερα δεν είναι, τόσο κοντά ε, στο αρχικό κείμενο που πολύ, ε, ήταν πολύ προσανατολισμένο προς τις ε, δημόσιες προμήθειες. Έχουμε πολλές λεπτομέρειες πρέπει να συζητήσουμε. Θα τις συζητήσουμε φαντάζομαι και εδώ στην Επιτροπή μας αλλά και με τους σκιώδεις εισηγητές και νομίζω ότι πλέον έχουμε ένα ισορροπημένο κείμενο. Μπορούν να το δεχθούν οι περισσότεροι. με ένας αμετανόητος αισιόδοξο άνθρωπος και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε εφιώς να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Τρίτο σημείο για τις τροπολογίες. Για πάρα πολλά σημεία αληθεύει ότι διαφέρουν σε κά... οι απόψει κάποιων συναδέλφων. Άλλοι θέλουν να είμαστε πολύ πιο αυστηροί σε σχέση με το κείμενο, άλλοι θέλουν να είμαστε πολύ πιο ευέλικτοι από το κείμενο. Και όλα αυτά συνεπάγονται εκ διαμέτρου αντίθετης απόψη, όπως καταλαβαίνετε. Και εκεί πλέον θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους οι συμβαστικές τροπολογίες. Το σώμα του σχεδίου έκθεσης ε, και στο μεγαλύτερο μέρος του στηρίζεται και μιλώ κυρίως για τα εξή στοιχεία. Πρώτα απ' όλα η ελευθερία θέλετε των δημόσιων αρχών να μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο διαχείρισης που επιθυμούν. Το είχαμε συζητήσει αν θυμάστε καλά αυτό το σημείο εδώ και θα ήθελα να είναι σαφές και στην έκθεση. Χαίρομαι λοιπόν που πολλοί συνάδελφοι έχουν υιοθετήσει σχετικές τροπολογίες και μάλιστα επεκτείνω ακόμα περισσότερο αυτή την πολύ σημαντική διάταξη. Επόμενο σημείο. Πολλοί από εμάς είμαστε ιδιαίτερα ε, ευνοϊκά δικαιωμένη στην μεγαλύτερη ελευθερία των δημόσιων αρχών που Πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφασίζουν τι κανόνα θα χρησιμοποιήσουν. Οι ίδιες δηλαδή οι αρχές θα πρέπει να αποφασίζουν για τους κανόνες που θα ε, εφαρμόσουν. Και βέβαια υπάρχουν οι γενικές αρχές της διαφάνειας, της ισότητας, της ε, ισότητας μεταχείρισης των υποψηφίων. Οι αρχές όμως είναι αυτές που θα πρέπει να αποφασίσουν για τους κανόνες και βέβαια μετά να εφαρμόσουν τους κανόνες που αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν. Αυτό έγινε αντικείμενο πάρα πολλών τροπολογιών, αλλά ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία. Επίσης, πώς μπορούμε να κάνουμε πιο ευέλικτο το είναι κάτι που ενδιαφέρει πολλούς συναδέλφους. Είμαι στο σημείο αυτό αρκετά αισιόδοξο ό,τι αφορά τους ορισμούς. Ιδίω στους κινδύνους, TST, παραχώρες κτλ. Έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες και σε αυτά τα σημεία και φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αφήσεις συμβιβασμούς. Δύο είναι τα βασικά σημεία είναι οι εξαιρέσει αρχής και οι τομεακές. Εκεί βέβαια πρέπει να δούμε από εκείνου κάποια πράγματα. Και το δεύτερο είναι η ενίσχυση των διατάξεων για κοινωνικές περιβαλλοντικές παραμέτρους. Πρέπει να σημειώσουμε πρόοδος προς αυτό το σημείο. Να δείξουμε μια συλλογική ευφία αν θέλετε. Τελευταίο σημείο και μετά κυρία Πρόεδρε γιατί μακρηγόρησα θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναντέλφους. Δύο τεχνικά ζητήματα για τις τροπολογίες. Για την τροπολογία 240, συγκεκριμένα απόρριψη της οδηγίας, η τροπολογία του ΕΛΚ είχε παρουσιαστεί ότι είναι, αλλά δεν είναι ακριβώς ε, έτσι τα πράγματα μαζί με την ΚΟΕ και τους Πρασίνους. Μάλλον έγινε ένα σφάλμα στην ε, κατάθεση της ε, τροπολογίας αυτής είναι συνάδελφοι καθόλου ε, αξιότιμοι, οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπούν το ΕΛΚ. θα πρέπει να γίνει μια διόρθωση εκεί και στην αγγλική έκδοση της ε, τροπολογίας 685 για τον υπολογισμό της αξίας παραχώρησης. Ε, είναι ένα σφάλμα λοιπόν. Στα γαλλικά, στην αρχική τροπολογία είναι σωστά Ουσιαστικά πρόκειται για επανάληψη τη 106 τροπολογία για το σχέδιο έκθεση. Δεν θα πρέπει πλέον δηλαδή να αναφέρεται το κόστο εκμετάλλευση, δεν πρέπει να λαμβάνετε υπόψη στην αξία τη παραχώρηση. Είναι μια πάρα πολύ συγκεκριμένη περίπτωση και σα παραπέμπω στην γαλλική έκδοση. Αυτή λοιπόν είναι αυτή που θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Ευχαριστώ. Vielen Dank für die Klarstellung und für Ihre Ausführungen. Ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση. Κύριος Παντσέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον ε, συγκεκριτή μας, τον κύριο Ζουβά, για την εισήγηση αυτή και για το νέο έγγραφο εργασίας που μας υπέβαλε. Είναι εξαιρετικό μέσο για να διευκολύνουμε τις διαπραγματεύσεις και να προωθηθούν οι τροπολογίες που έχουμε προτείνει. Να τον καθησυχάσω. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί μια θετική οδηγία που να οδηγήσει στην εναρμόνιση του ευρωπαϊκού, της ευρωπαϊκής αγοράς. Χωρίς να περάσω σε λεπτομέρειες για λόγους πίεσης χρόνου, να σχολιάσω τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και πιστεύω ότι μπορούν να συνδυαστούν με τη συλλογιστική του εισηγητή ώστε να απλουστευτεί γενικότερα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η νέα, ο νέος ορισμός ε, των ε, συμβάσεων παραχώρησης και των υπηρεσιών είναι και σαφέστερες και αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τον πραγματικό οικονομικό κίνδυνο. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε εδώ την προθυμία του εισηγητή να δει και τις δικές μας θέσεις. Για τη διοικητική λειτουργία των δημόσιων αρχών, η δυνατότητα των αρχών αυτών να αποφασίζουν για την ε, διαχείριση και την εκτέλεση εργών αλλά και υπηρεσιών είναι σημαντικό στοιχείο. Όμως πρέπει να τονιστεί ότι απότερος σκοπός θέλουμε να είναι, ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και βιωσιμότητας. Ισότητα μεταχείρισης και προώθηση της οικουμενικής πρόσβασης, της καθολικής πρόσβασης της ε, δημόσιας καθώς και η προστασία της αρχής διαφάνειας για τις δημόσιες αρχές. Η δημοσιοποίηση και η διαφάνεια είναι στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στη συλλογιστική του εισηγητή, ώστε να υπάρχει συστηματική αξιολόγηση της λειτουργίας των δημοσίων αρχών και η δημοσίευσή της στο κοινό. Για το γενικό οικονομικό συμφέρον, εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι η οδηγία αυτή θα πρέπει να τονώσει την ελευθερία των δημοσίων αρχών ώστε να ορίζουν το πλαίσιο των υπηρεσιών καθώς και τους τρόπους χρηματοδότησης των ε, υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Τώρα για τα κοινωνικά και για τις οικονομικές πάνω για τα οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Θεωρούμε αυτή την πτυχή πολύ σημαντική και πιστεύουμε ότι η οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει την περιβαλλοντική και κοινωνική νομοθεσία όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την εθνική νομοθεσία και από τις συλλογικέ συμβάσεις, όπου πολλές φορές εκεί λαμβάνουν χώρα οι παραχωρήσεις, οι σύμβασεις παραχώρησης, όμως τα περιβαλλοντικά κριτήρια έχουν ε, περιληφθεί και λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και ε, άλλα κριτήρια στα κεφάλαια για την ε, κρίση και την αξιολόγηση των συμμετεχόντων, των υποψηφίων. Τώρα, για, την, για τον υποδιαγωνισμό θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια ε, η κανονική λειτουργία όλης της αλυσίδας ε, διοργάνωσης στους δημόσιους διαγωνισμούς, στις δημόσιες Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Ζημά για την προθυμία του να συζητήσουμε τι δικέ μα ιδέε και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμβαστικέ λύσει με τρόπο επικοδομητικό και πρόσφορο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παντσέρη. Κύριε Μπόζε, Μπουζόη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ξανευχαριστήσω τον κύριο Ζουβάν για την ε, έκθεση του. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ήταν εύκολο το έργο του, γιατί ήταν, ε, θα είναι και πολλές τροπολογίες που θα συζητήσουμε τις προσεχείς εβδομάδες. Δεν προλαβαίνω τώρα να συζητήσω όλες τις τροπολογίες, δεν είναι άλλωστε ούτε καν αυτός ο στόχος της σημερινή συζήτησης. Απλώς πολύ σύντομα να εξηγήσω ποια θέματα θα μας απασχολήσουν περισσότερο στις επόμενες συζητήσεις. Οι εξαιρέσεις είναι σημαντικές εδώ, ιδίως με τις τροπολογίες που αναφέρονται στις εξαιρέσεις, διότι σε κάποια κράτη-μέλη η παροχή κάποιων υπηρεσιών ε, σχετίζονται με συγκεκριμένους φορείς μην ξεχνάμε όμω ότι σκοπό τη νομοθετική αυτή πρόταση είναι ακριβώ να υπάρχει περισσότερο ανταγωνισμό και περισσότερη αξία για τα χρήματα που δαπανούν οι δημόσιε αρχέ, αλλά και περισσότερη ποιότητα υπηρεσιών για του φορολογουμένου. Ο αποκλεισμό κάποιων ε, συμβάσεων παραχώρηση που απευθύνονται σε ιδιωτικέ εταιρείε, το εδάφιο 11.3 χρήζει ε, διευκρινήσεων για τις εξαιρέσεις in-house θα πρέπει, τις κάθετες αυτές εξαιρέσεις, θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον ε, μπορεί να καλύπτονται και οι συμβάσεις που δεν ε, είναι συμβάσεις των δημοσίων αρχών. Στι κάθετε εξαιρέσει, το άρθρο 15 πρέπει να υπάρξει περιορισμό του στο ελάχιστο ώστε να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμό. Η εξαίρεση θα πρέπει να παρέχεται εκεί που η παραχώρηση δίνεται σε νομικό πρόσωπο ή σε συμβάλλουσε αρχέ ή φορεί, εφόσον αυτοί λειτουργούν στην ε, ενιαία αγορά. Ιδάλω, θα υπάρχουν στρεβλώσει του ανταγωνισμού γιατί για το εναπομέναν 10% των δραστηριοτήτων θα υπάρχουν στην αγορά εταιρείε στις οποίες δεν θα μπορεί να δοθεί καμία σύμβαση ε, και έτσι θα υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αλλά το 10% αυτό εξαρτάται και από τη λειτουργία του φορέα. Τώρα για την κάθετη εξαίρεση θα πρέπει και στην παράγραφο 15.2 να διαγραφεί η διάταξη αυτή. Διότι αντίκεινται στη λογική τις γενικότερες πρότασεις οι εξαιρέσεις αυτές. Το ίδιο και για τις παραχωρήσεις που ελέγχονται από κοινό από δύο περισσότερες συμβάλλουσες ε, αρχές ή φορείς. Δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε ως γνώμονα την μία ε, ελέγχουσα αρχή, διότι δεν είναι ε, η ευθύνη μόνον της ε, ελέγχουσας αρχής που μπορεί να ελέγχει τις δικές της υπηρεσίες και τμήματα, αλλά πολλές φορές μπορεί να υπάρχει κοινή ευθύνη. Η συνεργασία αυτή μπορεί να έχει στόχο να εκπληρώνει η ίδια δημόσια αρμοδιότητα. Και βεβαίω ε, η σωστή λειτουργία στην ε, κοινή αγορά. Τώρα για τη διάρκεια των παραχωρήσεων. Οι συμβάσει παραχωρήσεων είναι μια άλλη καθοριστική παράμετρος αυτής της οδηγία και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η διάρκεια των παραχωρήσεων θα πρέπει να περιορίζονται στο χρονικό διάστημα που χρειάζεται ένας ε, φορέας ώστε να αποσβέσει τα κόστη της λειτουργίας και της επένδυσης και να πληρώσει τους στόχου που ορίζονται από την αρχική σύμβαση, κυρίως τους στόχου των επιδόσεων. Να ολοκληρώσω ε, λέγοντα κάποια πράγματα για τι προθεσμίε υποβολή προσφορά και τη δυνατότητα τροποποίηση ε, ισχυουσών ε, συμβάσεων. Βάσει των κριτηρίων για συμμετοχή στον διαγωνισμό θα συμφωνήσω με τα άρθρα 37 και 38 όπως έχει προτείνει να διατυπωθούν ο εισηγητή ο κ. Ζουδά. Όμω το όριο των 30 ημερών για τόσο περίπλοκε προσφορέ είναι πολύ σύντομο. Υπάρχει πρόβλημα με νέε προσφορέ που θα... δεν θα διευκολυνθούν καθόλου με τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό αντίκειται στο γενικότερο στόχο του νομοθετήματος. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι καλύτερα να έχουμε 52 ημέρες όπως αρχικά είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλος, για την τροποποίηση των συμβάσεων παραχώρησης. Όπως έχει υποθεί, σε πολλές περιπτώσεις οι συμβάσεις είναι πολλές φορές ημιτελής ή μακράς διαρκείας. Οπότε απαιτείται ευελιξία στην διάρκεια κατά την οποία ισχύουν. Θα πρέπει όμως η τροποποίηση αυτή να οριστεί βάσει αυτηρών κριτηρίων ώστε να μην υπάρχουν ε, στρεβλώσεις ή καταχρήσεις ανάλογα με τη φύση του σύμβαση και εφόσον αυτή δεν επηρεάζεται, η τροποποίηση θα, μπορεί να επιτρέπεται, θα μπορούσε να επιτρέπεται, αλλά μόνο εφόσον είναι επί τη ουσία και εφόσον προβλέπεται ω δυνατότητα στην αρχική σύμβαση. Και εφόσον βέβαια και η αξία τη τροποποίηση είναι κάτω από το 15% τη συνολική αξία τη σύμβαση. 5% προτείνει ο εισηγητή. Μου φαίνεται πολύ μικρό για μια σύμβαση παραχωρητική. δεδομένου του χαρακτήρα των συμβάσεων αυτών. Και ελπίζω βεβαίω ότι συζητώντα το αυτό με του συναδέλφου θα καταλήξουμε σε συμβαστικέ λύσει. Σα ευχαριστώ πολύ για το έργο σα και ανυπομονώ να ξανασυνεργαστούμε για αυτή την πολύ δύσκολη και περίπλοκη νομοθετική πρόταση. Και με τον κύριο Ζιβάν και με του υπόλοιπου συναδέλφου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρούλε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να καταστήσω Σαφέ, ξεκινώντα ότι δεν έχω διαβάσει σε κάθε λεπτομέρεια την τελευταία τροπολογία, αλλά πάντως θα ήθελα να πω ότι βλέπω ένα ευρύ φάσμα θέσεων να καταγράφεται από τις προτάσεις των ε, ομάδων. Ένα πρόβλημα που διαβλέπω ωστόσο έχει να κάνει με τη στοχοθέτηση αυτής της οδηγίας και μάλλον χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιλέξει αν θέλει διαφάνεια περισσότερο ή άνοιγμα στις αγορές. Ε, έχω την εντύπωση ότι από διαφορετικέ τοποθετήσει των πολιτικών ομάδων ε, ακούγονται διαφορετικά θέματα και διαφορετικέ τοποθετήσει, δηλαδή για πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τίνω να συμπεράνω ότι μάλλον θέλει να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου. Από την άλλη ωστόσο έχει τοποθετηθεί ρητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέρ του ανοίγματο αγορά μέσα από την οδηγία αυτή. Άρα λοιπόν ε, ίσω θα πρέπει να είναι πιο στενοί οι ορισμοί εδώ, πιο αυστηρές διατάξεις, έτσι ώστε να ε, γίνει το άνοιγμα των αγορών υπό πιο ελεγχόμενες συνθήκες. Αυτό όμως θέλουμε εν τέλει. Είμαστε εμείς εκείνοι μέσα στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπαθούμε να έχουμε στο δυνατόν πιο μεγάλη ελευθερία και τα κράτη-μέλη ώστε αυτά να αποφασίζουν εν τέλει πώς θέλουν να λειτουργήσουν όλα αυτά. Μια ακόμη παρατήρηση και νομίζω ότι και ο κύριος Μπουσόη συμφωνεί με, την υπο... με το άνοιγμα της αγοράς. Πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν ε, και να ορίσουμε πάνω απ' όλα τι θέλουμε με την οδηγία αυτή, τι επιδιώκουμε να επιτύχουμε την οδηγία αυτή. Κάτι πολύ σημαντικό εν προκειμένου είναι αυτό με το θέμα της ελευθερίας το οποίο τοποθετηθήκατε πολύ ωραία. Αλλά υπάρχουν και προτάσεις της ε, σοσιαλιστικής ομάδας οι οποίες Δίνω την εντύπωση ότι μάλλον για περιοριστικές συνθήκες, ε, μάλλον τείνουν να εισαγάγουν περιοριστικές συνθήκες όπως στην περίπτωση των δημόσιων προμηθειών στις υπηρεσίες. Αν είναι έτσι, ωστόσο, ε, περιορίζουμε πάρα πολύ το πεδίο ε, δράσης των φορέων ε, των ε, επιχειρήσεων και έτσι δεν θα έχουμε καλή υπηρεσία για τον καταναλωτή. Καλό θα ήταν λοιπόν να προσδιορίσουμε καταρχάς αυτό που μας είχε εξ αρχής υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια οδηγία light, θα λέγαμε ένα ε, πλαίσιο ελαφρύ που θα λειτουργήσει απρόσκοπτα. Άκουσα λοιπόν και τι θέσει των ομάδων, έχω ακούσει και τι θέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι το καλύτερο για το Κοινοβούλιο θα ήταν να απορρίψει την πρόταση στο βαθμό που αυτή δεν μπορεί να μα προσφέρει ασφάλεια δικαίου, αλλά μάλλον το αντίθετο. Και όσο δεν προσδιορίζεται επακριβώ, τι επιδιώκουμε. Θέλουμε άνοιγμα τη αγορά ή θέλουμε μόνο να αποφύγουμε τι προσφυλιέ στα δικαστήριο. Γιατί η θελουμε μονο να αποφυγουμε τι προσφυγε στα δικαστηρια γιατι η ασαφεια ως προς τη στοχοθέτηση μπορεί να σημάνει και το άνοιγμα των ασκών του αιώλου και να συνοδευτεί από, αμέριστες, ε, από αμέτρητες προσφυγές στα δικαστήρια και δικαστικές διαφορές που ασφαλώς δεν είναι προς το συμφέρον μας. Άρα λοιπόν ούτε τηρογημένες είναι αυτές τις θέσεις, ούτε βλέπω να προσφέρουν τίποτα επιπλέον. Η κυρία Βάιλερ, ευχαριστώ. Από το ECR είναι κανείς εδώ παρόν. Όχι, η Γκουε, ούτε. Η ΕΦΤ, ούτε. Επομένως, θα ακούσουμε τώρα πρόσθετες παρεμβάσεις Βάιλερ, Σφάπ και ΒΑΙΣΚΑΙΛΕΡ. Εγώ ήθελα να διατυπώσω μια ερώτηση προς τον εισηγητή, τον κύριο Ζουβά, ή και την Επιτροπή ενδεχομένω. Γιατί ομολογώ ότι ενοχλήθηκα όταν άκουσα τον κύριο Μπουζόη να μιλάει για τις ε, για την ανάγκη να περιοριστούν οι συνθήκες και οι όροι για τις ε, παραχωρήσεις και το λέω αυτό ξεκάθαρα. Ε, καταρχάς στη Γερμανία υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις. Ε, πάντως πιστεύω ότι ο κύριος Ζιβό, αλλά και πολλοί σοδημοκράτες, αλλά και άλλοι συνάδελφοι και εγώ επιμένουμε ότι θέλουμε λαμβάνεται η, απόφαση από τις δημόσιες αρχές εκεί όπου πρέπει να ληφθεί η απόφαση στην κάθε περιοχή, στην κάθε χώρα και αντιστοίχως να μπορεί να κριθεί από το δικαστήριο εάν υπάρχει πρόβλημα σε μια περίπτωση όπου για τρία-τέσσερα χρόνια δεν έχουν ληφθεί τέτοιες αποφάσεις. Όχι λοιπόν αυτό το οποίο ο κύριος ε, Μπουζόη μόλις πρότεινε, δηλαδή πολύ στενά όρια και περιορισμούς. Κύριε Μπουζόη, κύριε Ζουβέν, συγγνώμη, εσείς μπορείτε τουλάχιστον να τοποθετηθείτε προς τη διεύρυνση μάλλον, προς την πιο ευέλικτη ε, λύση ή το αντίθετο. Ο κύριος Φαπ πρώτα, μετά η κυρία Βάζικερπερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει. Προφανώς δεν έχουμε διαβάσει όλοι τις τροπολογίες των πάντων. Και ούτε εγώ βέβαια μπορώ να ισχυριστώ κάτι τέτοιο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ τον κύριο Ζουβάν γιατί έδειξε πνεύμα συνεργασίας και συμβασμού πολλά από αυτά τα οποία είχαμε προκαταβολικά ζητήσει ε, τα βλέπουμε εγγεγραμμένα μέσα στην έκθεση, ως βάση συζήτησης δηλαδή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχουν απαλληφθεί όλα τα προβλήματα. Πάντως, βλέπω να ακολουθεί ένα καλό δρόμο, ένα σωστό δρόμο προς την απλούστευση. Στο άρθρο 11, στην απλουστευμένη δυνατότητα, για τις ε, κοινοτικές, κοινοτικά οργανωμένες ε, δραστηριότητες. Βλέπω ότι υπάρχουν προτάσεις, αλλά θα ήθελα καταβολικά να επισημάνω ότι έχουμε αναθέσει τρεις μελέτες για να εξετάσουμε λίγο περισσότερο την αιτιολόγηση, τη βάση καλύτερα αυτής της οδηγίας, το λόγο ύπαρξης Είχα την ευκαιρία τις προηγούμενες ημέρες ε, στην Πράσινη Εβδομάδα χωρίς συνεδριάσει να μελετήσω αυτές τις ε, μελέτες και πρέπει να πω ότι προβληματίστηκα, άλλωστε το ε, κοινοποίησα και στο Policy Department, στο σχετικό τμήμα μελετών. Πρέπει να πω λοιπόν ότι είναι περίπλοκες οι συνθήκες και σε, σε κάθε κράτος μέλος ισχύουν πολύ διαφορετικές συνθήκες, όχι μόνο προς το νομικό πλαίσιο, αλλά και ως προς τις πολιτικές ή διοικητικές παραδόσεις που ισχύουν και θα είναι μάλλον αδύνατο να βρεθεί μια κοινή λύση, ένα κοινό παρονομαστής. Είναι πολλά τα προβλήματα, όπως επεσήμανε και η κυρία ε, Ρούλε νωρίτερα. Ε, τώρα, στο άρθρο 11 λοιπόν μιλήσαμε. Επίσης θα ήθελα να πω ότι κατά τη συζήτηση οδηγία, δεν θα πρέπει και να λησμονούμε ότι όπως άλλωστε πολλές φορές έχει υπογραμμίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει ασάφεια δικαίου, είναι ασαφείς οι συνθήκες και οι διατάξεις. Το είπε και ο συγκητής ίσως να θέλει κάτι να προσθέσει ακόμη μετά. Είναι κάτι που σύστησαμε την προηγούμενη εβδομάδα και στην ίδια του την ε, κοινότητα, την ιδιαίτερη πατρίδα, υπήρξε μια παραχώρηση η οποία έγινε τελικά αντικείμενο διορθώσεως ως προς την ευρωπαϊκή διάσταση. Πολλές αντίστοιχες συμβάσεις νομίζω θα υπάρχουν και άρα χρειάζεται διευκρίνηση των διατάξεων χωρίς να θέλω όμως να τοποθετηθώ οριστικά προς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει αυτό. Πάντως, πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε ένα κοινό παρονομαστή εάν εισαγάγουμε περισσότερη ευελιξία μέσα στη διαδικασία αυτή, η οποία εν τέλει σημαίνει ταυτόχρονα και ότι δεν θα ρυθμίσουμε 100% τα πάντα. Και ε, έχοντας πει αυτό, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρέπει πολιτικά να λαμβάνετε, πρέπει και πολιτικά να λαμβάνετε βεβαίω η απόφαση για την κάθε προσφορά, αλλά θα πρέπει και το κοινό τότε να είναι σε θέση να κρίνει, να ενημερωθεί για ποιο λόγο ποιο επικράτησε η μία προσφορά αντί της άλλης. Έτσι λοιπόν, να μην κοιτάμε μόνο κριτήρια ανταγωνισμού, αλλά και άλλα κριτήρια, αλλά να μπορούμε να τα βλέπουμε με κάποιο τρόπο πρέπει αυτά να εισαγάγουμε στο κείμενο, αλλά πιστεύω εν γέννη και κλείνοντα ότι ο κύριο Σουβέν έχει βρει μια σωστή κατεύθυνση με την του. Η κυρία Βάη Κέρμπερ, ευχαριστώ πολύ. Και καταρχά ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Ζουβά για την καλή συνεργασία. Θα θέλω να αναφερθώ σε κάποια σημεία εκφράζοντας και την πεποίθησή μου ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία και επικοδομητική σχέση. Θα ήθελα να πω καταρχά ότι συμμερίζομαι τις θέσει τη κυρίας ε, Ρούλε. Και νομίζω πολλοί είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι δεν είναι ακόμη αναγνωρίσιμη η προσθέμενη αξία της εκθέσεως, τη οδηγίας καλύτερα. Και διερωτώ με, γιατί η οδηγία αυτή χρειάζεται. οι παραχώρηση, οι παραχώρησης ε, έχουν ε, υπερσυνοριοκό χαρακτήρα, γιατί πρέπει να έχουμε λοιπόν πανευρωπαϊκή ρύθμιση. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν οδηγευτή. Εάν παρόλα αυτά, ωστόσο, η πλειονότητα των συναδέλφων τοποθετηθεί υπέρ τη εισαγωγή μια οδηγία στο πεδίο αυτό, θα ήθελα να διορθωθούν κάποια σημεία, σημαντικά σημεία, έτσι ώστε και να αποφευχθεί η υπερβολική γραφειοκρατία, αλλά και να εξασφαλιστεί επαρκή ευελιξία για τι ε, κοινότητε, για του Δήμου, αλλά όχι μόνο και για αυτού, και για μικρότερε και μεσαίε επιχειρήσει, τι οποίε λέμε ότι δηλώνουμε ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε. Αλλά νομίζω ότι δεν το έχουμε καταφέρει. Για τα επιμέρους σημεία λοιπόν, ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω και να υποστηρίξω τόσο είπε η κυρία Βάιλερ ως προς την ε, συνεργασία μεταξύ κοινοτήτων στις παραχωρήσεις. Νομίζω ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον ε, αναφέρονται σε δημόσιες δραστηριότητες, σε δημόσιες παραχωρήσεις, σε δημόσιες συμβάσεις, πρέπει να συμπληρωθούν από οδηγίες από διατύπωση μάλλον μέσα στην οδηγία, γιατί αυτή που έχουμε μέχρι τώρα δεν είναι επαρκής, δεν καλύπτει δηλαδή τη δυνατότητα που ενδεχομένω να ήθελαν αρκετοί δήμοι να συνεργάζονται μεταξύ τους. Αυτό το βλέπουμε στα δημόσια έργα στις πόλεις στη Γερμανία. Υπάρχει ένα μοντέλο ε, εργασίας εκτέλεσης των έργων, το οποίο είναι ικανοποιητικό, το οποίο θέλουμε να διαφυλαχθεί και το οποίο κινδυνεύει και λόγω της οδηγίας για, τις, ε, για την παροχή των υπηρεσιών αλλά και για την ε, οδηγία για τις παραχωρήσεις εδώ, να μην λειτουργήσει ικανοποιητικά. Γι' αυτό παρακαλώ να γίνει σχετική διόρθωση στην, ε, στις διατάξεις των δύο αυτών οδηγιών. Επίσης έχουμε την ε, παθητική συμμετοχή κεφαλαίου, ιδιωτικού κεφαλαίου. Όσο αυτό δεν είναι καθοριστικής σημασίας, το ιδιωτικό κεφάλαιο, τότε θα πρέπει να ακολουθήσουμε την νομολογία του δικαστηρίου. Και δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε σε υποχρεωτική ε, διαδικασία διαγωνισμού εφόσον δεν είναι κατά κύριο λόγο ιδιωτικό το κεφάλαιο το οποίο αναμειγνύεται στην σύμβαση αυτή, στην σύμβαση παραχώρησης. Το ποσοστό επίσης θα μπορούσαμε να το ξανασυζητήσουμε. Γιατί νομίζω θα πρέπει να αφορά μόνο δραστηριότητες που έχουν ουσιώδη σημασία για την εκτέλεση του έργου και όχι περιθωριακή σημασία. Νομίζω ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε το κείμενο περαιτέρω για να, βρούμε καλά, για να βγάλουμε καλά αποτελέσματα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι στις ε, παραχωρήσεις πρέπει και έχουμε καταθέσει τις σχετικές ε, τροπολογίες γιατί δεν υπάρχουν διεθνείς δεσμεύσεις ως προς το δίκαιο των παραχωρήσεων άρα δεν ισχύει το σχετικό επιχείρημα Μπορούμε να βρούμε λοιπόν νομίζω συμβαστικές λύσεις και ίσως θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε για άλλη μια φορά τις ε, εξαιρέσεις ή παρεκκλήσεις γιατί ο κύριος Σουφέ έχει εξαιρέσει κάποιους τομείς αλλά όχι κάποιους άλλους. Ας είμαστε λοιπόν συνεπείς και ας πούμε εφόσον κάποιος τομέας εξαιρείται ή κάποιοι τομείς εξαιρούνται τότε ίσως και οι άλλοι, φεριπίν, διάσωση, φεριπίν, τομέας των υδάτων θα πρέπει και αυτοί να ε, συμπεριληφθούν ε, ή να εξαιρεθούν καλύτερα το ίδιο και στον τομέα της ενέργειας. Στον τομέα των υδάτων είναι ξεκάθαρο το συμφέρον ε, της υγιεινής, ε, της προστασίας της δημόσιας υγείας κτλ. Όλα αυτά πρέπει να τα κοιτάξουμε πολύ μεγάλη προσοχή γιατί και η ιδιωτικοποίηση του τομέα των, ε, της σύντρευσης ενέχει πάρα πολύ σοβαρούς κινδύνους. Το ίδιο και στις υπηρεσίες διάσωσης. Εγώ που προέρχομαι από παιδιάδα, ξέρω πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει επαρκής ε, ρύθμιση έτσι ώστε όταν στην Ήπεθρο, όταν δεν ε, υπάρχει επαρκής απόδοση ή κερδοφορία από δραστηριότητες διάσωσης, να εξασφαλίζεται η εγκατάσταση η λειτουργία ενός δικτύου ικανοποιητικού στην Ήπεθρο, επαναλαμβάνω, χωρίς ε, να χρειάζεται να παρεμβαίνουμε. Επομένως, θα ήθελα να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και ε, κλείνω υπογραμμίζοντας ότι θεωρώ ότι η οδηγία καν χρειάζεται. Κυρία Βάιλερ, πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή οτι θεωρω οτι η οδηγια αυτη ουτε καν χρειαζεται Κύριε βαιλερ πριν δωσω το λογο στην ευρωπαικη επιτροπη Για την κυρία Βάισκερπερ, θα ήθελα να πω σύντομα ότι παραθέσατε τι δικέ μου θέσει και είπατε ότι συμφωνείτε, αλλά εγώ θα έλεγα, θα υπογράμμιζα καταρχά ότι θεωρώ ότι για λόγου ακριβώ ασφάλεια δικαίου είναι απαραίτητη αυτή η οδηγία. Μια σειρά από υπηρεσίε όμω, όπω αυτέ των υπηρεσιών διάσωση, θα πρέπει να είναι δυνατόν να οργανωθούν με διαφορετικό τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ σημαντικό να τοποθετηθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας μιλήσει για τις οριακές τιμές, είναι διαφορετικές από αυτές τις εκθέσεις του κυρίου Τεραβέλα. να μας μιλήσει για τις εξαιρεσει. Ναι, και ο κύριος Σουβέ ίσως θέλει στο τέλος να συνοψίσει ε, τοποθετούμενος όμως και ως προς τα ποσοστά που ε, μας ανέφερε η κυρία Βάισκερπερ. 90, 80, 85% τι ποσοστά θα προτιμούσατε εσείς. Γιατί υπάρχουν διαφορετικέ προτάσεις. Βλέπω τον κύριο Μάγερ όμως, ο οποίος το λάβει το λόγο πριν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να λάβω το λόγο πριν να μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, νομίζω ότι η νομοθεσία μπορούμε να εισάγουμε όταν έχουμε αρμοδιότητα, όταν είναι δυνατόν δηλαδή κάτι τέτοιο. Μπορούμε να κάνουμε επίση νομοθεσία όταν έχει νόημα, όταν είναι λογική η εισαγωγή μιας αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να εισάγεται ένα νομοθέτημα όταν είναι απαραίτητο. Αυτά, αυτούς τους τρεις όρους λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε και αν δούμε την, ε, τις αναφορές στον τύπο την προηγούμενη εβδομάδα στη Γερμανία αλλά και σε άλλα κράτη, τότε μάλλον καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι όλο και πιο επιφυλακτικοί, επιφυλακτικοί οι πολίτες ε, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως αυτό έχει να κάνει και με, την, ε, με τη, ε, ταμείο διάσωση και όλα αυτά τα μέτρα που εισάγονται και την κρίση και λοιπά ω συνήθω. Αλλά, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί ο πολίτη να ξεχωρίσει τι είναι εθνική αρμοδιότητα, τι είναι ευρωπαϊκό δίκαιο. Τι κάνουν οι Ευρωπαίοι, τι κάνουν οι εθνικέ κυβερνήσει. Όπω παραδείγματι με το πακέτο διάσωση. Έτσι λοιπόν, με το Ταμείο Διάσωση. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για νομοθεσία εκεί όπου πράγματι φέρνει κάποια αλλαγή ουσιαστική στη ζωή των ανθρώπων. Όταν η νομοθεσία είναι τέτοια η οποία επιβαρύνει, ώστε να επιβαρύνει τον ε, πολίτη με κόστος υψηλό, γραφειοκρατικό, για να κάνει τη δουλειά του σε κάτι τόσο πάρα πολύ απλό, όπως βλέπουμε καμιά φορά να συμβαίνει, τότε είναι απαράδεκτο να την νομοθεσία. Και εδώ Θεωρώ ότι, είναι απα... ότι πρώτον η νομοθεσία αυτή δεν είναι απαραίτητη, πρώτο επιχείρημα. Δεύτερο επιχείρημα είναι σε ένα βαθμό, σε ένα βαθμό μόνο έχει νόημα η εισαγωγή της, μικρό βαθμό, όχι εν γέννη και όχι συνολικά έχει νόημα. Όπως είπα λοιπόν, σε ορισμένα μέρη της έχει νόημα αυτή η οδηγία, ε, αλλά θεωρώ ότι το να έχει νόημα ε, μερικώς δεν αρκεί. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε ένα νέο νομοθέτημα δεν ε, σημαίνει ότι υποχρεωτικά πρέπει και να το πράξουμε. Και έτσι, κυρίε και κύριοι, έχουμε εδώ μια πρόταση, έχουμε έναν συγγητή, έχουμε τον κύριο Ζουβέ, τον αγαπητό και αξιότιμο συνάδελφο, τον φυσικά, ε, για τον οποίο δεν έχω καμιά προσωπική ε, επιφύλαξη. Απλώ θεωρώ ότι το νομοθέτημα αυτό πραγματικά δεν χρειάζεται και θα πρέπει να εξετάζουμε και να μελετάμε τι θέλουμε, τι χρειάζεται να κάνουμε και αν δεν είναι απαραίτητο κάτι να το κάνουμε, να μην το κάνουμε. Και πάνω απ' όλα αν δεν έχει νόημα. Αυτό τα λέω με ένα κάπως έντονο ύφο, το, τα συγγνώμη, διότι πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ειδικά αυτές τις εποχές, ώστε ό,τι μέτρα να λαμβάνουμε να έχουν και νόημα και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω για τις τροπολογίες που μας στείλατε και για τις προσπάθειες ε, και το έργο που επιτελεί η Επιτροπή σας για τις μας παραχώρησης. Ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα την όλη προσπάθεια παρά τις δυσκολίες και τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα του εν λόγω νομοθετήματος. Όπως έχουμε είπε και κατά το παρελθόν, Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το σχέδιο έκθεσης του εισηγητού και με τις λύσεις που προσφέρει το έγγραφο αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την εξέβρεση μιας καλής λύσης για ένα θέμα που χρήζει ρυθμίσεις και θα επανέλθω σε αυτό. Το κείμενο λοιπόν ε, γίνεται πιο ξεκάθαρο, πιο απλό και αυτό είναι μια καλή βάση εργασίας. Μπορούμε λοιπόν να προσυπογράψουμε το σχέδιο εκθέση του εισηγητού. Βέβαια, οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί είναι πολυάριθμες και πηγαίνουν σε διάφορες κατευθύνσεις. Δεν μπορώ βέβαια να επεκταθώ στην καθεμία χωριστά. Θα κάνω κάποια γενικά σχόλια για ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για αυτή την οδηγία. Επίσης όμως θα ήθελα να απαντήσω στους ισχυρισμούς περί σύγχυσης για το στόχο της οδηγίας. Νομίζω ότι κατέστη ξεκάθαρο ότι αρχικά αυτό που προσφέρει η οδηγία αυτή είναι ένα εργαλείο για τις ε, δημόσιες προμήθειες, δηλαδή αγορές ε, που κάνουν δημόσιες αρχές με, δημόσια, με δημόσιους πόρους. Δηλαδή, έχουμε κανόνες για τις δημόσιες ε, προμήθειες εδώ και 40 χρόνια, αλλά όχι για τις παραχωρήσεις. Έχουμε συμβάσεις έργους συμβάσεις υπηρεσιών παρόμοια είναι τα πράγματα. Βέβαια υπάρχουν κάποιε ιδιαιτερότητε και για αυτέ προσφέρονται συγκεκριμένε λύσει. Αλλά αυτό για το οποίο συζητούμε σήμερα είναι τα εργαλεία για αυτέ τι δημόσιε προμήθειες. Η οδηγία αυτή, υπό την έννοια αυτή, προσφέρει πρόσβαση και στι οικονομικέ δραστηριότητε για όλου του παράγοντε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε για την εσωτερική αγορά, για τι δημόσιε προμήθειε. Επομένω, όλοι οι οικονομικοί παράγοντε, Γερμανοί, Πολωνοί, Φιλανδοί, οτιδήποτε, Βρετανοί, έχουν απόλυτο δικαίωμα στο να έχουν πρόσβαση στη δραστηριότητα αυτή όταν παρέχεται αλλού, ακόμη και το ίδιο βέβαια ισχύει για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και θα πρέπει να δούμε πώ θα μπορέσει να τι βοηθήσει περισσότερο αυτή η οδηγία. Τι βοηθάει λοιπόν τι μικρομεσαίε προσφέροντά του πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα. Πρόθεση τη οδηγία λοιπόν είναι οι κανόνε να είναι στο δυνατόν πιο απλοί. Με σειρά προτεραιότητα λοιπόν. Είναι ένα εργαλείο για τι δημόσιε προμήθειε, παρέχει πρόσβαση σε όλου του οικονομικού παράγοντε και με τον απλούστερο δυνατό τρόπο. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, δέσμευση των τροπολογιών. Πρώτη, περί απόρριψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη με τις τροπολογίες αυτές, αλλά κατανοούμε ότι είναι και ένα ενδεχόμενο. Χαιρετίζουμε πάντως το γεγονό ότι η προθυμία είναι να υπάρξει επεξεργασία κάποιων πτυχών αυτή τη οδηγία και η απόρριψη απλά είναι μία επιλογή. Είναι μία από τι φωνέ που ακούγονται. Πάλι διευκρίνηση ό,τι αφορά το στόχο, το σκοπό. Υπάρχουν και τροπολογίες για την ε, ε, περαιτέρω αποσαφήνιση του στόχου. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική των υπηρεσιών, εμείς αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο είναι χρήσιμε τροπολογίε σχετικέ, αλλά και τροπολογίε που μιλούν για τι υπηρεσίε γενικού οικονομικού ενδιαφέροντο, που επαναλαμβάνουν την ελευθερία που έχουν οι δημόσιε αρχέ να οργανώνουν τι εν λόγω υπηρεσίε με τον τρόπο που επιθυμούν. Καλοδεχούμενε και οι δύο σχετικέ διευκρινήσει. Ό,τι αφορά τι εξαιρέσει τώρα, αν η οδηγία αυτή θέλουμε να έχει κάποιο νόημα, θα πρέπει να έχει και κάποιο αντικείμενο. Οι τροπολογίε λοιπόν που ε, προτείνουν να εξαιρεθούν όλες οι υπηρεσίες οικονομικού ε, συμφέροντος και μη, θα έλεγα ότι ουσιαστικά πηγαίνουν και ενάντια στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συνομοθετούν, είναι προφανέ αυτό, αλλά πολύ ξεκάθαρα το Δικαστήριο λέει ότι καλύπτονται οι υπηρεσίε οικονομικού ενδιαφέρου από του κανόνε των δημοσίων προμηθειών. Η εξαίρεση λοιπόν τομέων, με άλλα λόγια, που καλύπτονται από τι υπηρεσίε αυτέ, είναι κατά τη νομοθεσία, κατά τη νομολογία του δικαστηρίου. Σε ό,τι αφορά τι υπηρεσίε μη οικονομικού ενδιαφέροντο, εκεί ξεκάθαρα λέγεται ότι μπορεί να μην εφαρμόζονται για τι υπηρεσίε αυτέ οι κανόνε περί ανταγωνισμού, εφαρμόζονται όμω οι κανόνε περί δημόσιων προμηθειών. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε τι υπηρεσίε, τι είδου υπηρεσίε ε, ε, αφορά αυτή η οδηγία. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διασαφήνιση του τι είναι ή δεν είναι παραχώρηση, και αυτέ οι τροπολογίε είναι χρήσιμε, γιατί καλό είναι να είναι ξεκάθαρα και οι εγκρίσει και οι που δεν καλύπτονται. Και οι σχετικέ τροπολογίε λοιπόν είναι χρήσιμε τώρα. Για το public public operation. Το ανέφεραν πολλοί ομιλητέ. Η πρόταση πράγματι, όπω ε, έχει υποβληθεί από την Κομισιόν, ουσιαστικά ε, ακολουθεί την ομολογία. Κάποιε πτυχέ όμω ε, πηγαίνουν λίγο πιο μακριά και προσφέρουν μεγαλύτερη δυνατότητα δημόσια-δημόσια συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να παρέχεται η ελευθερία αυτή στις δημόσιες αρχές. Εξού και διατυπώθηκαν έτσι στο άρθρο 15 οι σχετικές διατάξεις. Προσοχή όμως γιατί το δικαστήριο αναφέρεται ρητά σε συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών. Άρα οποιαδήποτε συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου θα πρέπει να αποκλείεται. Αυτή είναι και η λογική, είναι το λογικό επακόλουθο. Όταν έχουμε δηλαδή αμυγός μια in-house situation, ε, κάθετη κατάσταση, δεν υπάρχει τους κανόνες. Τώρα, για τις, τρο... για τις τροποποιήσεις. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια εξέλιξη των σχετικών συμβάσεων και πάντοτε βέβαια τηρώντας τη νομολογία. Είναι χρήσιμη λοιπόν η λύση σε ό,τι αφορά τη διάρκεια ζωής της σύμβασης παραχώρησης και ένα τελευταίο γενικό σχόλιο αριθμός τροπολογιών δηλαδή σε σχέση με τις προτάσεις ε, των κρατών μελών και του Συμβουλίου. Ήδη υπάρχει αρκετή σύγκληση σήμερα, δηλαδή και τα κρατημέλη και οι προτάσεις ορισμένων τροπολογιών πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Και έτσι όλα αυτά ε, συνηγορούν στο να έχουμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση και στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κυρία έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είμαι σίγουρη ότι καταλάβατε, ότι απαντήσατε στην ερώτησή μου για τις οριακές τιμές. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, κυρία Ρουλέ, Πρόεδρε, επιτρέψτε να ρωτήσω το εξή. Λέτε ότι η ερμηνεία του γενικού συμφέροντος υπάγεται στη σχετική νομολογία του δικαστηρίου για την ε, νομοθεσία αυτή. Νομίζω ότι είναι πολύ ευρύ αυτή η ερμηνεία και αν διαβάσει κανεί την ε, συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η έννοια του δημοσίου συμφέροντο ανήκει μόνο στα κράτη-μέλη κατά αρμοδιότητα και, μεικτή, και συντρέχουσα αρμοδιότητα έχουμε μόνο για τι οικονομικέ υπηρεσίε. Η Επίτροπη. Ευχαριστώ πολύ. Για τι υπηρεσίε Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είδε την πρόταση στι τροπολογίε που εξηγούν ότι η διοργάνωση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντο ω τομέα του, του, των κρατών μελών είναι και σημαντικό και πολύ απαραίτητο. Κάτι που συμβαίνει και με την ισχύουσα νομοθεσία. Όμω πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η εξαίρεση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντο από το πεδίο τη οδηγία δεν είναι κάτι που το θεωρεί εφικτό το δικαστήριο. Ότι υπάρχουν πολλέ υποθέσει που έχουν εξεταστεί από το ΔΕΚ και ακριβώ ασχολούνται με τι υπηρεσίε γενικού οικονομικού ενδιαφέροντο. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι το Eurobus, η υπόθεση αυτή. Και όσον αφορά τα ανώτατα όρια, η κατάσταση διαφέρει ελαφρώς σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις, αλλά όχι και πλήρως. Δηλαδή, δεν υπάρχει απόλυτη ελευθερία στο να ορίζονται τα ανώτερα επίπεδα, διότι υπάρχουν δύο διμερείς ε, διεθνείς συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, με ε, ορισμό του ε, επίπεδου των ανώτερων όριων. Εάν θέλουμε να διαπραγματευτούμε διαφορετικά τα ανώτατα όρια, θα υπάρξουν συγκεκριμένε συνέπειε σε διεθνέ επίπεδο. Δεν υπάρχει λοιπόν κάλυψη DPA, αλλά υπάρχουν δύο διμερεί συμφωνίε για, το... για το επίπεδο των ανώτατων ορίων και πόσο μπορούν να εγωριστούν. Ναι, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, κυρία Ρίλε. Το ερώτημα ήταν εάν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτές τις διμερείς ε, συμβάσεις. Ε, ναι, λέει η κυρία Βάιλερ και εγώ. Ήθελα να παρακαλέσω γραπτός να ενημερωθούμε για τι συμβάσει. Τι συμβάσει εννοείται ακριβώ. Και έχουμε την τάση εδώ στην Επιτροπή μας να ε, αυξάνουμε τα όρια, τι οριακέ τιμέ, αφετέρου δε να είμαστε προσεκτικοί στις ε, συναλλαγέ με τις τρίτες χώρες. Γι' αυτό παρακαλώ λοιπόν όταν έχετε τα στοιχεία να μα τα αποστείλετε. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει το λόγο. Έχουμε εξαντλήσει νομίζω το θέμα. Παρακαλώ τον κύριο Σουβά. Για να κλείσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κράτησα πυροτοδός ε, σημειώσεις από τη συζήτηση. Ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω σε όλα. Καταρχάς, μια παρατήρηση για τον Χάνς Πίτερ. Πάντοτε είναι πολύ επιτυχημένο να ακούει κανείς ε, ότι όταν η Ευρώπη ασχολείται με όλα τα πάντα πάνε καλά όμως. Εδώ θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου είδου δηλώσεις διότι επιτυχίες μπορούμε να έχουμε στην κοινή γνώμη λέγοντας ε, κάνοντας τέτοιες δηλώσεις αλλά δεν πρέπει αυτή την ευκολία να τη χρησιμοποιούμε. Είμαστε πολίτες ε, ευρωπαϊκού, του ευρωπαϊκού έθνους, οικοδομούμε ένα νέο έθνος με μια συλλογική προσπάθεια και με τρόπο έστω βραδύ πρέπει να υιοθετήσουμε κοινού κανόνες. Είμαστε, και αυτό είναι η δουλειά μας, είμαστε υπεύθυνοι για να δημιουργήσουμε το νομοθετικό σώμα. Να επιτρέψουμε να προχωρήσει η συλλογική θεώρηση των πραγμάτων. Το δικό μου ιδανικό είναι μια Ευρώπη όπου αύριο, έστω και μεθαύριο, θα συμφωνήσω εδώ μαζί σα, θα μπορούσαν να υπάρχουν κοινοί κανόνε από το βορρά στο νότο τη Ευρώπη. Το να λέμε ότι η Ευρώπη κάνει υπερβολικά πολλά, μακάρι, αυτό έχω να πω, μακάρι να ομογενοποιούσε τα πράγματα η Ευρώπη και να γίνονταν όλα κοινά. Θα ήταν πάρα πολύ καλό. Τέλο πάντων, για να απαντήσω στην κυρία Βάιλερ με ρωτήσατε την φιλοσοφία που υποκινεί την έκθεση μου, δηλαδή πέραν των τεχνικών τροπολογιών, το τι πιστεύω. Κατά πρώτον, η παραχώρηση είναι ένα εργαλείο και μόνον. Ένα πρόσθετο εργαλείο που δίνουμε στις δημόσιες αρχές. Έτσι πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Επίσης πρέπει να επαγρυπνούμε ώστε η παραχώρηση να μην γίνει ένας, μια μέθοδος ιδιωτικοποίησης ε, από την πίσω πόρτα. Όχι, είναι ένα εργαλείο που δίνουμε στις δημόσιες αρχές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή και όχι. Τελεία εκεί όμως. Δεν πρέπει να αρχίσει η συζήτηση για το αν είναι καλύτερο να ιδιωτικοποιηθεί διαχείριση των υδάτων ή όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν έχω απάντηση. Απλώς θα ήθελα οι δήμαρχοι οι νομάρχες, οι πρόεδροι των επιφερειών, να μπορούν να αποφασίσουν με τους υπόλοιπους ερετούς εάν ε, θα διαχειριστούν ε, το... τη συγκεκριμένη υπηρεσία με αυτόν τον τρόπο ή όχι. Δηλαδή in-house ή όχι. Εάν επίσης θέλουν να έχουν αυτή την προσωρινή διαχείριση, αυτόν τον προσωρινό τρόπο διαχείρισης. Δηλαδή να αναθέσουν σε ιδιωτικό φορέα προσωρινά την ε, διαχείριση αυτή. Και πράγματι, επιτρέψτε μου εδώ και μια παρέκβαση. Διότι υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το κείμενο δεν είναι καλό, επειδή ακριβώ θα είναι για την πόρτα στι ιδιωτικοποίησει. Αυτοί που τα ισχυρίζονται αυτά υπερασπίζονται ένα σύστημα, ακούστε με εδώ, ένα σύστημα όπου στην ουσία ένα μέρος των δημοσίων υπηρεσιών ήδη ανατίθενται σε ιδιωτικού φορεί. Με συμβάσει απεριορίστου διαρκεία και με στρέβλωση του ανταγωνισμού. Επιτρέψτε μου, εγώ αυτό το ονομάζω ιδιωτικοποίηση. Με τέτοιε προποθέσει. Αυτό που ακριβώ θέλαμε λοιπόν είναι όταν πράττουμε κατά αυτόν τον τρόπο αυτό να γίνεται με διαφάνεια, με ίση μεταχείριση των υποψηφίων και με συνθήκες ε, αντικειμενικές. Εάν δούμε τώρα την ομολογία του 10 εδώ και 10 χρόνια σε σχέση με τις παραχωρήσεις, υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος υποθέσεων. Εδώ λοιπόν πρέπει να οικοδομήσουμε ένα ευρωπαϊκό έθνος, αυτό έλεγα προηγουμένως. Για να απαντήσω λοιπόν στη συνάδελφο, αντικειμενικά, οι παραχωρήσεις είναι διακρατικός τομέας. Παράδειγμα, η υπόθεση Κέλσεν Weiser, εταιρεία δημοσίου δικαίου, εκτός από το 1,3% του κεφαλαίου της. 1,3% ανήκει σε ιδιώτες. Το υπόλοιπο είναι δημόσιο περιουσιακό στοιχείο. Η εταιρεία αυτή συμμετέχει αυτή τη στιγμή σε διαγωνισμό για τη διαχείριση των υδάτων στην περιοχή του Μπορντό. Θα μου πείτε ότι το θέμα αυτό είναι λίγο αντιφατικό διαχείριση των υδάτων στον Μπορντό, διότι το Μπορντό είναι πιο γνωστό για τα κρασιά του παρά για τα νερά του. Παραμένει όμως ένα ζήτημα αντικειμενικό. Μην λέμε μεταξύ μας ότι δεν έχει διακρατικές διαστάσεις. Απλώς το νόημα που θα πρέπει να αποδώσουμε σε όλο αυτό το θέμα είναι το εξή. Κατά πόσον οι δημόσιες αρχές θέλουν να υπάρχει και συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου στη διαχείριση κάποιων υπηρεσιών. Ας γίνει αυτό. Αλλά ας γίνει με διαφάνεια. Αυτό λέμε. Να μην ε, υπάρξει αποκλεισμό επιλογών. Να υπάρχει ελευθερία επιλογή. Και το γνωρίζουμε και για ιστορικού λόγου αυτό. Όλε οι χώρε ε, εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Είναι περίπλοκο το θέμα αυτό. Κάποια πράγματα λειτουργούν και αναγκαζόμαστε να τα ισοπεδώνουμε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο για να υπάρξει και εμπίστοση χρόνου πίστοση χρόνου για να μπορέσουν τα διάφορα συστήματα να προσαρμοστούν. Ένα παράδειγμα του οποίου εγώ ίδιο υπήρξα θύμα. Είμαι δήμαρχο μια κοινότητα κοντά στο Παρίσι. Το 2004 εμπιστεύτηκα σε εταιρεία κατά 70% ιδιωτικού κεφαλαίου ε, παραχώρηση, σύμβαση παραχώρηση στην κοινότητά μου. Ανέλαβαν τη διαχείριση κάποιου πράγματο, τέλο πάντων, κάτι χωροταξικό. Το 2004. Τον καιρό εκείνο δεν ε, είχαμε κάνει διαγωνισμό διότι υπήρξε ιστορικά ήταν ε, υπεύθυνο αυτό ο φορέα. Το 2012 έληξε βάσει απόφαση Γαλλικού Δικαστηρίου η παραχώρηση λόγω τη Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Και ξεκίνησαν, ε, ξεκίνησε διαγωνισμό. Τώρα μια σύμβαση 200 εκατομμυρίων ευρώ που λύγει ε, από τη μια μέρα στην άλλη, επειδή δεν έγιναν σεβαστέ οι βασικέ αρχέ του Ευρωπαϊκή συνθήκε, αυτό θα ευχόμουν να μην σα συμβεί σε κανέναν σα εδώ. Διότι πρέπει να σα πω πραγματικά τι σκέφτομαι. Και να το πω ξεκάθαρα. Νομίζω ότι κοροϊδεύουμε του εαυτού μα όλοι μαζί, εάν πιστεύουμε ότι εφόσον αυτό πάντα γινόταν, δεν θα αλλάξει κιόλα. Όχι, θα έρθει ένα δικαστή και θα πει αυτή η νομική δομή που διαχειρίζεται την τάδη υπηρεσία για την τάδε κοινότητα δεν ε, έχει σεβαστεί τις βασικές αρχές της συνθήκης, δεν έχει γίνει ανάθεση με διαφάνεια, οπότε πάβει η σύμβαση. Έρεται η νομιμότητα της, ε, του συγκεκριμένου φορέα τη εταιρεία. Αυτό συνέβη και σε εμά και για να μπορέσουμε να βγούμε από το αδιέξοδο θα πρέπει να αποφασίσουμε τι εξαιρείται και τι συμπεριλαμβάνεται. Ιδιωτικό κεφάλαιο. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός με απλές διαδικασίες πάναπλε. Αλλά να συμφωνήσω εδώ με την κυρία Ρίλε. Η διαδικασία είναι απλούστατη. Και δεδομένη η διαδικασία που εξηγραμε είναι μια διαδικασία που λέει το εξή. Δύο στάδια. Πρώτον, ως δημόσια αρχή δηλώνω ότι πρέπει να υπάρξει διαγωνισμό για το τάδε ζήτημα, για το τάδε αντικείμενο. Δηλώνω την πρόθεσή μου δηλαδή να υπάρξει διαγωνισμός και μετά δηλώνω τη διαδικασία επιλογής και κάνω αυτό που θέλω. Βάσει κανόνων βεβαίως που έχω υπαγορεύσει προηγουμένως. Αλλά μπορεί να γίνει τόσο απλά και αυτό αρκεί. αρκεί. Δεν είναι τόσο κοπιώδε. ούτε για τι δημόσιε αρχέ. Είναι απλώς μία εγγύηση. Εγγύηση ότι κάνουμε αυτό που επιδιώκουμε με τρόπο ισότιμο οι δημόσιες αρχές μπορεί να θέλουν να κρατήσουν οι ίδιες την ε, διαχείριση κάποιων υπηρεσιών, την υδροδότηση, την ηλεκτρική ενέργεια, τα απορρίμματα. Αν θέλουν ε, να παραμείνουν in-house αυτές οι υπηρεσίες, αυτές οι παραχωρήσεις, θα πρέπει να πούμε με σαφήνεια, πολύ ξεκάθαρα. Με να ρωτήσετε για το 10%, για το 20%, ποια είναι η φιλοσοφία μου. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι πραγματικοί αριθμοί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν καν. Η φιλοσοφία μου είναι η εξής ένα παράδειγμα πάλι. Μια δομή δημοσία, δημοσίου συμφέροντο. στο Παρίσι λόγου χάρη που ασχολείται με τη συγκομιδια απορριμματων απορριμμάτων. In-house, 100% δημόσια. Θα μπορούσε αύριο να πει θέλω τα, η συγκομιδή να ασχοληθεί με τη διαχείριση απορριμμάτων στο Στρασβούργο. Και συμμετέχω σε διαγωνισμό. Η... Το σημαντικό είναι το ποσοστό το ποσοστό που θα αναλάβει η πόλη του Παρισιόλογου χάρη, αν θα είναι 10%. Γι' αυτό ακριβώς ψάχνουμε τα ποσοστά, για να μην υπάρχει ψευδής ανταγωνισμός, τρέβλωση και για να ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν μιλάμε λοιπόν για ιδιωτικοποίηση, συνάδελφοι, ούτε αυτό επιδιώκουμε και πρέπει να επαγρυπνούμε. Και έπειτα οι δημόσιε αρχέ πρέπει να διατηρούν τα ημεία, Αυτοί να υπαγορεύουν του κανόνε. Τώρα, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κανόνε που έχουν υπαγορευτεί από τι δημόσιε αρχέ, θα πρέπει να ακολουθούνται από όλου. Και τέταρτον, εφόσον θέλουν να διαχειριστούν οι ίδιοι οι δημόσιε οι δημόσιε αρχέ τη υπηρεσία, α το κάνουν. Αλλά εφόσον υπάρχει διαγωνισμό, θα πρέπει να υπάρχει και κοινή λογική. Εφόσον μπορεί να γίνει επιλογή από πολιτικού άνδρε και γυναίκε, τότε να υπάρξει και διαγωνισμό ανταγωνισμό. Για να μην μα συμβούν τα δυσάρεστα, οι περιπέτειες που σα περιέγραψα και τι έχω ζήσει εγώ ίδιο. Από το 2004 ανατέθηκε αυτή η διαχείριση στην εταιρεία, στην εταιρεία που σα προανέφερα, αλλά όχι γιατί ήταν φίλοι ούτε ημέτεροι. Ιστορικά είχαν αναλάβει ε, αυτή τη διαχείριση και ήταν πολύ πιο απλό πραγματικά αν το ήξερα από, σήμερα, τι θα είχε, από τότε τι θα είχε συμβεί σήμερα, θα περίμενα άλλο ένα εξάμεινο, θα είχε γίνει μια δημόσια διαδικασία και τώρα δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Δεν θέλω εδώ να είμαι δογματιστή. Απλώ προσπαθώ να τραβήξω την προσοχή σα και να σα επισημάνω το εξή. σε κάποιες περιπτώσεις το δημόσιο κεφάλαιο και το ιδιωτικό είναι συνδεδεμένα και είναι δύσκολο να υπάρξει αντικειμενικός ανταγωνισμός όπως τον αντιλαμβανόμαστε. Σε μερικά χρόνια θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Και άλλοι Γάλλοι συνάδελφοι, θυμόμαστε πολύ καλά στη Γαλλία πριν από 25 χρόνια, όταν ε, εγκρίναμε παρόμοιου νόμου, με έναν μοναδικό σκοπό του εγκρίναμε. Να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Διότι γνωρίζουμε ότι κάποιες δημόσιες αρχές έκαναν τις επιλογές του τάδε ή του Βίνα για λόγους ευκολίας ε, σχέσεων. Αυτό ήταν ο στόχος εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω αν πρέπει να παραμείνει στόχος μας ακριβώς αυτό και σήμερα, αλλά αν μπορεί να εξυπηρετήσει σε κάτι, γιατί όχι. Πρόεδρε, αυτά είχα να πω. Ελπίζω να, μην, να ήταν αρκετά πλήρης η τοποθετήσή μου. Ähm, Ευχαριστώ. Και λεπτά. Ακόμα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς να ευχαριστήσω τον Φιλίπ για αυτά που μόλις είπε και να καθησυχάσω όσους αμφιβάλλουν και αισθάνονται βεβαιότητα. Η τελευταία φράση του Φιλίπ ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Στη Γαλλία, όντως, προηγουμένως τα πράγματα ήταν μια ζούγκλα είναι ένας από τους σπάνιους νόμους, ε, και εδώ πραγματικά είμαι αυστηρή, από τους σπανιότατους που κανείς δεν αμφισβήτησε και τελικά όλοι εκτιμούν, είτε τοπικές, περιφερειακές, δημόσιες αρχές και οι ιδιώτες. Συμφωνείς μαζί μου Φιλίπ, ήταν πραγματικά ένα άλμα, ένα άλμα διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και προστασίας ταυτόχρονα και των καταναλωτών και των δημοσίων πολιτικών τέλο πάντων αρχών και διοικητικών. Το είπα, δεν έχουμε εμεί διαφθορά στην υδροδότηση. Ε, μην φανταστείτε ότι δεν έχουμε υδροδότηση στη διαχείριση των υδάτων. Μάλλον δεν έχουμε διαφθορά στην υδροδότηση στη Γερμανία και έχετε μόνο στην Γαλλία και σε εμά συμβαίνει. Σα ευχαριστώ θερμά, κύριε Σουβά. Μια μικρή παρουσίαση. Σύντομη τοποθέτηση, αλλά και φιλοσοφική θα έλεγα. Συνάμα Κάτι το οποίο πρέπει όλοι μας να συμμεριστούμε, πιστεύω, να τοποθετούμε θα όλοι οι φιλοευρωπαϊστές κατά των επιθέσεων εις βάρος των, της Ευρώπης. Και επίσης μιλήσατε για την διαφθορά. Βεβαίως, μπορεί να μην έχουμε τέτοιου τύπου διαφθορά στη Γερμανία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαφθορά στις δημόσιες υπηρεσίες, στις δημόσιες αναθέσεις είχαμε περιπτώσεις και Γερμανών πολιτικών που βρέθηκαν ε, υπόδικοι. Και επίσης η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Crime ε, μόλις επιστρέφει από την Σικελία, όπου ξέρετε το ζήτημα της διαφθοράς είναι πολύ σημαντικό. Και στις ε, συμβάσεις παραχωρήσεως Άρα κάθε κράτος, όχι μόνο στον νότο της Ευρώπης, αλλά σε κάθε μέρος, πιστεύω, θα μπορούσε να επωφεληθεί από ένα. Η κυρία Ρούλε, χωρίς μικρόφωνο. Η πρόεδρος. Ναι, η διαφθορά έχει ενισχυθεί όντως και από την οικονομική κρίση σε ορισμένα κράτη. Πάντα θα υπάρξουν εκείνοι οι οποίοι θα έχουν την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα να αξιοποιήσουν μια δύσκολη κατάσταση σε ένα κράτο. Εάν εμεί όμω μπορέσουμε να βοηθήσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε απλέ, σαφεί δομέ, μπορούμε νομίζω να πούμε ότι έχουμε επιτελέσει το έργο μας, ότι η Ευρώπη έχει επιτελέσει το έργο της. Θα ήθελα να πω, κλείνοντας κύριο Σουβά, ότι προβλέπετε ψηφοφορία στις 18 Δεκεμβρίου, κύριε Ζουβά. Ψηφοφορία για την ε, σημαντική αυτή έκθεση με όλες τις συμβαστικές προτάσεις και τροπολογίες 18 Δεκεμβρίου. Το επαναλαμβάνω γιατί θα είναι η τελευταία μέρα από ό,τι φαίνεται που θα έχουμε βουλευτές στις Βρυξέλλες και γι' αυτό θέλω να είναι σαφές και για τους συντονιστές γιατί δεν αρκεί για ένα τόσο σημαντικό νομοθέτημα να έχουμε μόνο 5-6 βουλευτές παρόντες. Πρέπει οι συντονιστές να το σκεφτούν καλά εάν 17-18 του μηνός θα έχουμε αρκετούς βουλευτές. Εγώ εδώ θα είμαι, δεν υπάρχει θέμα, αλλά να προσέξουμε παρακαλώ, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Αυτό λοιπόν ήταν η έκθεση. Αυτή ήταν η έκθεση του κ. Ζουβέ για τι συμβάσει παραχώρηση και περνάω τώρα στο τελευταίο θέμα όπου βλέπω ότι ο εισηγητής και η Σκιώδης και ο Σέγγελ συγκεκριμένα δεν είναι ακόμα εδώ. Α, ο κύριος Φάπ θα τον αλάβει. Καλώς. Παρέχουμε τον Σκιώδη εισηγητή, αλλά ο εισηγητής ε, των σοσιαλδημοκρατών όπου να είναι θα φανεί από ό,τι φαίνεται. Να και ο κύριος Δεζόν, κύριε Ρούλη είναι εδώ. Δύο λεπτάκια διάλειμμα. Ο κύριο Τωραπέλα είναι στον δρόμο από ό,τι φαίνεται. Ε, liebe kolleginnen und kollegen liebe gäste liebe mitarbeiter αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι και συνεργάτες έχουμε ένα θέμα πολύ σημαντικό τώρα τα σημεία 7 και 8 συγκεκριμένα της σημερινής διάταξης του κυρίου Ταραμπέλα των Σοσιαλδημοκρατών για τις δημόσιες συμβάσεις. Κύριε Ταραμπέλα, έχετε το λόγο. Merci. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι διαπραγματεύσει για τι δημόσιε συμβάσει τι τελευταίε εβδομάδε σημείωσαν πρόοδο και οι πολιτικέ ομάδε έχουν συζητήσει ε, το ίμιση των κλάστερ, των δέσμεων, το 1 και το 4, δηλαδή δικασίε και procurement. Υπάρχουν βέβαια για το 3, 7, 8 και 2 κάποιες, ε, κάποια ανοιχτά ζητήματα και τα 5, 9, 10 κλάστερ δεν τα έχουμε ακόμη αγγίξει. Θα δούμε όμως το 9 και το 10 σήμερα. Σε ό,τι αφορά τώρα την αμοιβαιότητα, την διακυβέρνηση, την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, ε, είναι θέματα σημαντικά τα οποία θα τα αναφέρουμε σήμερα. Είναι χρήσιμη συζήτηση για να δούμε τι ε, πρεσβεύουν οι μεν και οι δε για τα ζητήματα αυτά και την πέμπτη θα τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω, Τετάρτη, Πέμπτη. Πέμπτη. Έχουμε την επόμενη συνεδρίαση των σκιωδών. Να ξεκινήσω λοιπόν με αυτό το οποίο συζητήσαμε το, με τους σκιώδεις, το 7 παραδείγματος χάρη κλάστερ για τη διαφάνεια και ιδίω τις ε, διάφορες παραλλαγές. Στόχος μας βέβαια είναι να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά αυτές τις μεταβλητές, που πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να είναι κάτι που επιτρέπεται αυτή εξ αρχή, γιατί έτσι μπορεί να έχουμε κάποιε δημοσιονομικέ ολιστήσει. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αυτό να το αναφέρει η προκήρυξη του διαγωνισμού και να μην έχει ως αποτέλεσμα αχρίαστο κόστος. Βελτίωση των διαδικασιών στο κλάστερ 8. Για μένα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της όλης οδηγίας και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του θέματος. Σύγκρουση συμφερόντων είναι ένας ορισμός που πρέπει να γίνει εφαρμοστέως αφού πρώτα οριστικοποιηθεί. Σύγκρουση συμφερόντων δεν θα πρέπει μόνο τα οικονομικά και γενιακά δημοσιονομικά ζητήματα και για τα συναισθηματικά συζητήσαμε. Ήταν ε, η αρχή πρόταση επιτροπής, αλλά εγώ ε, θεωρώ ότι διαφάνεια είναι σημαντικό πυλώνα της οδηγίας αυτής και ιδίως το άρθρο 18 διατάξει ό,τι αφορά το απόρριτο. Έχουμε λοιπόν μια συμβαστική τροπολία καταθέσεις που θεωρούμε ότι είναι ισορροπημένη. Η αναθέτουσα αρχή δεν θα πρέπει τις εμπιστευτικές πληροφορίες να τις αποκαλύπτει, θα πρέπει να σέβεται και την πραγματική ιδιοκτησία, αλλά απ' την άλλη υπάρχει δυνατότητα δημοσίευσης κάποιων στοιχείων της σύμβασης για να υπάρχει διαφάνεια και έλεγχος των διαδικασιών ανάθεσης. Είναι ανοιχτή η μέθοδος εργασίας, γίνεται μια ε, συζήτηση, θέλω να υπάρχει συζήτηση με όλες τις πολιτικές ομάδες, με όλους τους κοιόδης, αλλά όπως ε, θέλω να επιθυμίσω και με τους υπεύθυνου ε, για αυτό το θέμα από τις 7 επιτροπές που θα γνωμοδοτήσουν. Κάποιες μάλιστα έχουν ήδη γνωμοδοτήσει για αυτό το θέμα. Μέθοδος αυτή βέβαια θα μας οδηγήσει πιστεύω σε συμβιβασμούς που ήδη ορισμένους τους έχουμε και άλλους ελπίζω να έχουμε στο μέλλον. Μπορεί να προκύψουν και κάποιες παρανοήσεις που θα πρέπει να τις ξεκαθαρίσουμε. Ίσως να μην καταφέρουμε βέβαια πάντοτε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και να έχουμε απογοητεύσεις, όπως σε ό,τι αφορά το 69 άρθρο για πάρα πολύ χαμηλές προσφορές, τα χαμηλές προσφορές. Ξέρετε ότι πολλές φορές, με πολύ χαμηλές προσφορές, θα πρέπει όμως να, πρέπει να τις εντοπίσουμε, να τις ανοιχνεύουμε. Μέσω λοιπόν αυτών των προσφορών βλέπουμε προσφορές που οδηγούν σε ανάθεση σύμβασης που δημιουργεί προβλήματα σε επίπεδο της υλοποίησης της Και επομένως ο στόχος είναι να έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα για τη σύμβαση. Τα ποσοστά λοιπόν για να ανοιχνεύουμε τις ε, προσφορές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό είναι ένα εργαλείο. Μπορεί να μην είναι εντελώ ε, επαρκές, αλλά είναι απαραίτητο για να καταπολεμήσουμε το dumping που απειλεί τις συμβάσεις, τους διαγωνισμούς. Δεν μπορεί να το καταργήσουμε εντελώ ε, αυτό το στοιχείο, αλλά θέλουμε τουλάχιστον να το ελαχιστοποιήσουμε. Οι περισσότεροι συνάδελφοι όμως προτιμούν να μην αναφερόμαστε σε χάσματα, σε αποστάσεις, σε ε, διαφορές ποσοστών δηλαδή, σε σχέση με ένα μέσο όρο. Τίτλος 4 μας δίνει κάποια εργαλεία για τον έλεγχο των ε, δημόσιων συμβάσεων. Στην έκθεσή μου εγώ δίνω ιδιαίτερη σημασία στην διακυβέρνηση, στο governance. Αναγνωρίζω βέβαια ότι παρά την πρόταση ε, της Κομισιόν που δεν ορίζει συγκεκριμένα τον έλεγχο, θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη που δεν έχουν έλεγχο ε, μέσω συγκεκριμένου οργάνου θα πρέπει να θεσπίσουν ένα τέτοιο όργανο. και αν υπάρχουν αρχέ να μην δημιουργήσουμε νέε και επιβαρύνουμε τη διαδικασία και υπάρχουν και κάποια ομόσπονδα κράτη που στρέφουν προ την Πρόεδρο. Ομόσπονδα κράτη που δεν έχουν ένα εθνικό όργανο ε, ομοσπονδιακό, αλλά σίγουρα κάποιο περιφερειακό ή σε επίπεδο κρατηδίων για τη Γερμανία. Να μην ε, ανακαλύπτουμε ή δημιουργούμε νέε αρχέ εκεί που υπάρχουν, αλλά εκεί που δεν υπάρχουν, τι δημιουργήσουμε αυτέ τι αρχέ, γιατί είναι σημαντικό για την παρακολούθηση, για τον έλεγχο και τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων για όλες τις χώρες μέλη της Ένωσης. Πριν να περάσω τώρα στο πεδίο εφαρμογή και στους ορισμούς, θα συζητηθούν την Πέμπτη, θα ήθελα να έχω τη στήριξή σας για την τροπολογία που καταθέτω για το άρθρο 16. Στο κλάστερ 8 αναφέρομαι. Στόχος είναι πιο εύκολη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα μπορούν να ε, συνιστούν όμιλο, κοινοπραξία. Είναι καλέ πρακτικέ αυτέ, τι βλέπουμε στην Ιταλία για παράδειγμα για την υποβολή μιας προσφοράς ε, από έναν ενίο οικονομικό φορέα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει για να έχουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε διαγωνισμού να μπορούν να ε, δημιουργούν ε, μια κοινοπαραξία γιατί ίσω ξεχωριστά να μην μπορούσαν να αποβάλουν μια προσφορά και θα ήταν καλό να μπορούν να, τις, να χρησιμοποιούν το εργαλείο αυτό η ΜΜΕ και έχουμε πολύ θετικέ εμπειρίε σε διάφορε χώρε μέλη για το public public operation, παρότι έχουμε πολλές τροπολογίες, ε, ελπίζω να φτάσουμε σε συμβιβασμό, γιατί νομίζω ότι πιο πολλοί θέλουν να υπάρχει ελευθερία στα κράτη-μέλη, να υπάρχει βέβαια και η σοβασμός αρχή της επικουρικότητας, αλλά και στις τοπικές ε, αρχές. Εξαρτάται βέβαια από την αποκλειστική αρμοδιότητα. Πού έχει αποκλειστική αρμοδιότητα το κράτος μέλος. σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική κοινωνική προστασία, νομίζω πρέπει να εξαιρεθεί, μου φαίνεται σημαντικό, αλλά συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν που λέει ότι δεν θα πρέπει να έχουμε διάκριση υπηρεσιών Α και υπηρεσιών Β. Στην αρχική μου έκθεση το βλέπετε. Αυτό δηλαδή ελαφρυμένε διαδικασίε και κοινωνικέ υπηρεσίε. Αυτή η light, η ελαφρυμένη αυτή διαδικασία, σίγουρα θα προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία και διαφάνεια. Το να διακρίνουμε τώρα το τομέα σε α και β δεν είναι καλό. Δεν θα πρέπει να έχουμε ένα τέρμονο κατάλογο εξαιρέσεων που ουσιαστικά αυθαίρετα θα δημιουργεί αυτό το διαχωρισμό. Αφού έχουμε την εσωτερική αγορά, καλό θα ήταν να αρχίσουμε να δεχόμαστε κάποιους κοινούς κανόνες. Και τώρα βέβαια είμαι όλος αυτιά αγαπητοί συνάδελφοι ω προς ε, τις ερωτήσεις που θα έχετε να υποβάλλετε για τα κλάστερα αυτά. Για κάποια φαντάζομαι ότι αποδίδεται μεγαλύτερη συμμαχία, αλλά έχουμε και τα τελευταία πέντε, το 6 έως το 10 και φαντάζομαι ότι κάποια συνάδελφοι θα εστιάσουν περισσότερο σε ορισμένα εξ αυτών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Vielen Dank, Ευχαριστώ Μάρκ Ταραβέλα. Ο κύριος Σφαπ. Είναι εδώ. Τους ελεύθερου κανείς. Ο η κυρία Ριουλέ, τους πρασίνους. Ο κύριος Κιγιόν. ECR δεν βλέπω κανέναν. Ας ακούσουμε όμως τον κύριο Σφαπ και μετά την κυρία Ριουλέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, όπως και στις παραχωρήσεις και στο θέμα των δημοσίων συμβάσεων, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε προχωρήσει, είναι κάπως καλύτερη οργάνωση, πιο απλές οι δομές. Θα ήθελα ωστόσο να πω ξεκινώντα ότι παρακολουθούμε βέβαια τις, ε, τα σημεία στα οποία έχει διαρθρώσει ο κύριος ε, Ταραμπέλα, αλλά μας ξαφνιάζει το γεγονός ότι μιλάει για την ε, παροχή των υπηρεσιών, ενώ από τον τύπο και τις δηλώσεις στον τύπο στο Βέλγιο είχαμε αντιληφθεί διαφορετική τοποθέτηση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πω ότι ορισμένα ζητήματα ε, θα είναι δύσκολο ε, να περάσουν. Το πρόβλημα για μας είναι περισσότερο η ουσία όμως και όχι τι θα πει η κοινή γνώμη. Γι' αυτό λοιπόν όταν λέει ο κύριος Ταραμπέλο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την απελευθέρωση των ε, κοινωνικών υπηρεσιών, νομίζω ότι κάνουμε μάλλον κακό στην υπόθεση της Ευρώπης. Καταλαβαίνω ότι έκανε τις δηλώσεις του πριν από τις ευρωπαϊκές κοινοτικές εκλογές, αλλά είναι λαϊκισμός το να λέει κανείς πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Γι' αυτό λοιπόν θα κοιτάξουμε το έγγραφο επικριτικά και θα κοιτάξουμε αν μπορούμε να κάνουμε και τις σχετικές τροποποιήσεις. Ε, μία διαπίστωση ότι υπάρχει προσπάθεια εδώ να υποτιμηθεί η να απαξιωθεί καλύτερα η οδηγία, δεν θα ακολουθήσει η ομάδα μας αυτή την προσπάθεια. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν να εξασφαλίσουμε μία λύση η οποία θα δίνει την πιο καλή, την πιο φθηνή, την πιο αποτελεσματική προσφορά και βέβαια πάντα με την ε, τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, με λιγότερη γραφειοκρατία και όσο το δυνατόν περισσότερη ευελιξία για τις αρχές. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η κύρια ιδέα που μας καθοδηγεί, ε, τον κύριο Έγγελ και ο και εμάς, τους υπόλοιπους, στη δουλειά μας και θα ήθελα να πω ότι με ό,τι διατυπώσει στην πρόταση πρέπει να είναι σε θέση όλοι οι συνάδελφοι να ε, συμμετάσχουν. Και συνεχίζω τώρα στα γαλλικά, γιατί μια και το έχω συζητήσει με τον κύριο Έγγελ στα γαλλικά, ε, θα ήθελα να διαβάσω το κείμενό του. Η ομάδα μας λοιπόν διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσει ορισμένα σημεία, αλλά υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές και συγκεκριμένα δεν θέλουμε το κείμενο αυτό να παρεκτραπεί του στόχου του για να αφαιρέσει ε, από τις δημόσιες αρχές το δικαίωμα ή μάλλον την ε, εξουσία για την... Ε, Κύριε Σφάπ, <laughs> λίγο πιο σιγά παρακαλούμε. Ε, του αντίον είμαστε διατεθειμένοι να εξηγήσουμε σαφέστατα ότι όλοι οι οικονομικοί παράγοντες θα πρέπει να σέβονται τα κοινωνικά δικαιώματα σε όποια χώρα δραστηριοποιούνται στο βαθμό που αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με άλλη υφιστάμενη στην Ευρώπη νομοθεσία και δει την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Εν τέλει παραμένει λίγος χρόνος μέχρι την ψηφοφορία. Ο κύριος Έγγελ, λοιπόν, ο συνάδελφος, ενθαρρύνει τον εισηγητή να καταθέσει τροπολογίες οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα στις ε, περισσότερες πολιτικές ομάδες ε, να τις επεξεργαστούν. Γιατί μέχρι τώρα οι συμβασμοί ήταν πολύ περιορισμένοι ως προς τις παραχώρησεις που προσέφεραν οι σοσιαλιστές. Προς το συμφέρον λοιπόν των πάντων θα μπορέσουμε να εργαστούμε εφόσον υπάρχει συμβασμό. Ιδάλλως θα χρειαστεί να καταφύγουμε σε ψηφοφορίε μεγάλου αριθμού τροπολογιών, μία προς μία. Και τώρα στα γερμανικά, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω στο 8 και το 9, τα σημεία 8 και 9 στο κείμενο και συγκεκριμένα στο άρθρο 15 με τις προτάσεις του κυρίου Ταραμπέλα. Για να πω ότι εμείς θα θέλαμε μια διατύπωση η οποία να είναι σύμφωνη με την αρχή περί αποσπάσεως, με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και με τις δημόσιες προμήθειες ε, και τη διατύπωση αυτή αν μου επιτρέπετε να σας τη διαβάσω, στα αγγλικά αυτή τη φορά όμως, αργά-αργά. Οι οικονομικοί φορεί θα πρέπει να προσαρμόζονται στην οικονομική, κοινωνική, εργατική νομοθεσία ως προς την απόσπαση υπηρεσιών και εργατικού δυναμικού όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Εθνικό Δίκαιο και να σέφονται όπου υφίστανται συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο και οικουμενικής εφαρμογή και αρχές οικουμενικής εφαρμογής. Εδώ λοιπόν έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με τα όσα προτείνει ο κύριος Ταραμπέλα. Πιστεύουμε όμως εμείς ότι πρέπει να είναι επαρκές, ε, είναι επαρκής η αναφορά στο ευρωπαϊκό δίκαιο, να, να είναι δηλαδή κατηφυντήρια... να είναι ο μήτρος Αριάδνη στο ευρωπαϊκό δίκαιο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μπορεί να ισχύει μια τη διάταξη λοιπόν στο βαθμό που είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε μια κατάσταση δύσκολη για την Ευρώπη οικονομικά νομίζω ότι μπορεί να φανεί αυτό κάπως δύσπεπτο αλλά πρέπει να το δεχθούμε γιατί αυτό είναι το σωστό. Επίσης, μια λογική λύση για τις παραχωρήσεις μπορεί να εξευρεθεί. Δεν θέλουμε εμείς μεγάλες κεντρικές δομές, ε, γιγαντιές δομές, αλλά μπορούμε με απλές δομές, και το έχει επισημάνει και ο κύριος Ταραμπέλα, και νομίζω ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν μέσα επικοινωνία, δίευλοι επικοινωνίας και ενημέρωσης που μπορούν να συντονιστούν και αυτή τη δουλειά μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κυκλοφορευτεί η ενημέρωση και οι πληροφορίες. Οι αρχές βεβαίως που θα θεσπιστούν θα πρέπει να είναι ε, τέτοιες ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα υπερβολικής γραφειοκρατίας στα κράτη-μέλη κτλ. Και αν μου επιτρέπετε τώρα, κυρία Πρόεδρε, θα δώσω την, ε, θα δώσω γραπτό βέβαια τι προτάσει στον κύριο Ταραμπέλα, αλλά θα σταματήσω εδώ για να αφήσω και του συναδέλφου να τοποθετηθούν. Περιμένω να ακούσω με πολύ ενδιαφέρον τι θέσει του. Η κυρία Βάιλερ. Ε, ναι, πριν ε, δώσω το λόγο στην κυρία Ρούλε, θα παρακαλέσω τον κύριο Σφαπ να δώσει τα κείμενα, το κείμενο του κύριου Έγγελ ε, στη γραμματεία μας έτσι ώστε να το διαβάσουμε εμείς τον κύριο Ταραμπέλα και τους λοιπούς σκιώδες ηγητές και βέβαια να έχουν την ευκαιρία να κοιτάξουν την πρόταση αυτή προσεκτικά, όπως είχαμε κάνει και με τον κύριο Κομφεράτη, η κυρία Ρούλα. Βλέπω ότι είναι και ο κύριος Κρόετσμαν εδώ, ίσως ε, είναι δυνατό να μιλήσει και εκείνο αργότερα. Πάντω, εγώ ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία. Αλλά έχουμε το εξή πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Στην Επιτροπή είχαμε πει ότι ένα από τα μια από τις κεντρικές δυσκολίες ω προς τις δημόσιες προμήθειες ήταν ακριβώς ότι έχει καταστεί πολύ περίπλοκος όλος ο τομέας, χωρίς αυτό να είναι ευθύνη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά περισσότερο του τρόπου με τον οποίο υλοποιείται αυτή στα, στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, αλλά και στα δικαστήρια. Έτσι λοιπόν, ο τομέας των ε, δημοσίων συμβάσεων είναι πολύ περίπλοκο. Στόχος μας είναι να τον, να τον απλοποιήσουμε, να τον απογραφειοκρατικοποιήσουμε και ούτω καθεξής. Ε, πολλές λεπτομέρειες όμως έχουμε συζητήσει χωρίς να κριθεί στις συνεδριάσεις των σχεδόν εισηγητών το κεντρικό αυτό ζήτημα της απλούστευσης της νομοθεσίας. Ε, εάν δεν λυθεί όμως ε, αυτό και το ζήτημα πάνω απ' όλα του γραφειοκρατικού φόρτου, γιατί όπως είπα είναι από αυτά που δεν έχουν επιληθεί, θα χρειαστεί η ομάδα μου να καταψηφίσει τι προτάσει. Προτείνω λοιπόν ε, να το ξανασυζητήσουμε. Βεβαίως και είμαστε υπέρ ε, της ιδέας μιας πιο φθηνής ε, πρότασης. Αυτή θα πρέπει να επιλέγεται, αλλά δεν θέλω να παραμείνει μέσα στο κείμενο ρητά αυτή η παραπομπή, αυτή η διάταξη περί φθηνής πρότασης, διότι θέλουμε εκτός από φθηνή η πρόταση να είναι και η πιο καλή και δεν θέλουμε η αναθέτουσα αρχή να βρεθεί σε μια κατάσταση όπου θα είναι αναγκασμένη να παραπέμπει στο δικαστήριο, να ζητάει ε, κρίση από το δικαστήριο και χωρί αυτή την κρίση του δικαστηρίου να μένει σε θέση να λάβει απόφαση. Αν λοιπόν παραμείνει αυτή η ιδέα τη ε, φθηνότερη λύση, θα οδηγηθούμε σε αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν και σας συνιστώ να ρωτήσετε και τις τοπικές ή δημοτικές αρχές της ε, πατρίδας σας, γιατί θα δείτε ότι ακριβώς αυτά τα προβλήματα θα έχουν και βέβαια το ζήτημα της ασφάλειας δικαίου είναι πάρα πολύ καθοριστική σημασία. Τώρα, στην νομοθεσία αυτή υπάρχουν κάποιες ε, έννοιες, κάποιοι όροι που χρησιμοποιούνται χωρίς να είναι ε, σαφείς, χωρίς να έχουν ξεκαθαριστεί δηλαδή από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να του αποφύγουμε. Αυτή είναι μια άλλη μεγάλη δυσκολία που βλέπω. Δηλαδή χρειαζόμαστε σαφείς ορισμού, σαφείς έννοιες, απλές έννοιες για να μην ε, είναι επιματέωλη αυτή η προσπάθεια και η αναθεώρηση. Ε, επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σε υπηρεσίες Α και Β, τις Β τις έχει καταργήσει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά αν αυτό είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, γιατί θέλουμε τώρα ευελιξία υποτίθεται. Και γι' αυτό λόγο δεν αντιλαμβάνομαι γιατί μας λέτε ότι αυτές ε, οι υπηρεσίες πλέον δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Νομίζω ότι θα πρέπει να τις ξανασυζητήσουμε και ιδιαίτερα τις υπηρεσίες, ε, τις υπηρεσίες Β και να δούμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται και τι είδους χαρακτήρα έχουμε. Ε, πέραν ε, των κοινωνικών υπηρεσιών, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και στις νομικές υπηρεσίες. Φανταστείτε μια επιχείρηση, καλύτερα μάλλον ένα δήμο ή μια κοινότητα η οποία θέλει να αναθέσει σε μια νομική επιχείρηση, ε, σε μια νομική εταιρεία την εκπροσώπησή της θα πρέπει να καταφεύγει σε διαγωνισμό ανά την Ευρώπη. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μια σαφής διακρίση μεταξύ υπηρεσιών Α και Β για να μπορούμε να διευκολύνουμε αυτή την ανάθεση και την εξασφάλιση των απαιτούμενων ε, υπηρεσιών χωρίς να χρειάζεται πάντοτε να γίνεται διαχωρισμός από την αρχή. Ένα πιο απλουστευμένο, πιο ε, ευέλικτο σύστημα δηλαδή. Αυτή η ευελιξία είναι ε, ανάγκη να εισαχθεί ταχύτατα και σε σχέση με αυτό που υπόθηκε νωρίτερα, οι μικρέ και μισέ επιχειρήσει ε, πάντοτε υπογραμμίζουν, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον από την εμπειρία μου, ότι θέλουν να έχουν στο δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε συγκεκριμένα το θέμα αυτό και αναλόγως να ψηφίσουμε. Νομίζω ότι οι λέξεις δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία όσο η ουσία. Για δε τι λογικέ ε, συμφωνίε ε, και τι παρατηρήσει του κυρίου Σφάπ, ήθελα να πω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με κράτη όπω την Νορβηγία, όπω η Ελβετία. Και εγώ έχω επικοινωνήσει την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα από το Στρασβούργο. Είχα ε, επικοινωνία και αλληλογραφία με την, με την Νορβηγία και με αντίστοιχε υπηρεσίε, οι οποίε μου λένε ότι κινδυνεύουν να μην σε θέση για λόγου συλλογικών συμβάσεων να συμμετάσχουν. Επομένω, όταν λέτε universally applicable ε, οικουμενικής εφαρμογής, κριτήρια ή αρχές οικουμενικής εφαρμογής. Δεν ξέρω αυτό τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει. Κινδυνεύουμε πάλι να εξαρτώμεθα από τις δικαστικές συμβάσεις ή ε, τις δικαστικές αποφάσεις. Δυστυχώς να χρειάζεται κάθε φορά να ερμηνεύουμε, να, να προς τα κάτω την, ε, τις απαιτήσει μας και τα κριτήριά μας. Ίσως πρέπει πρώτα να γίνει μια αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση για να εξασφαλιστεί διαφάνεια προς την υπόθεση αυτή, γιατί ασφαλώς υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία προσδιορίζουν ε, την, ε, τα τιμολόγια, τους μισθούς, ε, τα ημερομίσθια με βάση τις συλλογικές συμβάσεις, ενώ κάποια άλλα όχι. Και άρα θα πρέπει να βρούμε μια διατύπωση η οποία θα επιτρέπει σε κράτη όπως τα σκανδιναβικά ή η Νορβηγία Φερρυπίν να συμμετέχουν χωρίς προβλήματα στις διαδικασίες. <laughs> Yeah, Σας ευχαριστώ. Κύριε Κρότσμαν, εσείς. Also, ob wir das hinkriegen mit der Vereinfachung, äh, habe ich so meine Zweifel. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είμαι σίγουρη ότι διευκολύνουμε το στόχο της ε, πλούστευσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει στις ε, δημόσιες προμήθειες να έχουμε όσο το δυνατόν, δημόσιες συμβάσεις να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ε, ανοιχτό πεδίο δράσης, γιατί όσο πιο πολλά πράγματα ρυθμίζουμε, τόσο πιο ασαφής και αβέβαιη γίνεται η κατάσταση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, ένας δήμος ή κοινότητα θέλησε κάποια στιγμή να εγκαταστήσει ε, σωληνώσεις αποχέτευση που θα έπρεπε να περάνε από το δρόμο μπροστά από κάθε σπίτι για να ε, φεύγουν τα νερά των αποχετεύσεων. Αλλά από το δημόσιο διαγωνισμό που έγινε και από τις προτάσεις που κατατέθηκαν, βγήκε ότι θα ήταν σκοπιμότερο αντί να αντικατασταθούν οι υφιστάμενε σωληνώσει, να αγνοηθούν, να ε, σκαφτεί ο δρόμο στη μέση του και έχει πια στην άκρη προ το σπίτι κάτω από το πεζοδρόμιο, στη μέση του και εκεί να κατασταθούν νέες ε, για την αποχέτευση. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε σε ένα παράδειγμα πολύ ενδιαφέρον για το τι, πού μπορούμε να οδηγηθούμε αν κοιτάμε μόνο το, την πιο φτηνή λύση. Ε, επίσης ε, για τις ε, συμφωνίες πλαισίου και τη χρονική τους διάρκεια. Βεβαίως να το δούμε κυρία Ρούλη, αλλά τέσσερα χρόνια ίσως δεν είναι αρκετός χρόνος, μάλλον έξι είναι καλύτερα. Οι πληστηριασμοί επίσης, ε, οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί είναι ενδιαφέρουσα λύση, αλλά όχι πάντοτε η μόνη. Και να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, ότι μπορεί ε, στο χώρο πάλι των δημών και των να έχουμε περίπτωση όπου θεωρούν ότι είναι καλύτερη η ιστορική ανάθεση, ενώ για άλλο έργο να είναι πιο αποτελεσματική διαδικασία του διαγωνισμού. Επομένω, δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση που θα ισχύει για τα πάντα. Πρέπει να αφήνουμε ένα περιθώριο για ε, διερεύνηση διαφορετικών λύσεων ανα, περίπτωση. Όπως είπαμε, η πιο φθηνή λύση δεν είναι πάντα η καλύτερη. Ίσως, ίσως εάν εμείνουμε στην πιο φθηνή λύση θα πρέπει να πιέσουμε να εισαχθεί αυτό που ονομάζεται γερμανική ε, λύση, δηλαδή να εξηγείται κάθε φορά σε ποιο βαθμό είναι πιο φθηνή η λύση. Και πάνω απ' όλα διαφάνεια βέβαια, ώστε να είναι σαφή η όροι υπό τους οποίους ε, επιλέγεται μία ε, προσφορά. Και η αξιολόγηση του κόστου θα πρέπει να καλυπτεί όλους τους τομείς και τους, κοσ... και τους κοινωνικούς και τον οικονομικό τομέα και όλους τους άλλους και το περιβάλλον ακόμη. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ε, ε, ε, συμβάσεις οι οποίες δεν είναι τόσο καθαρές. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι να υπάρχει διαφάνεια όπως είπα και νωρίτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια. Και αιτιολόγηση της αποφάσεως. Είτε είναι η σύμβαση σχετικά ε, ε, η σύμβαση η πιο φθηνή λύση, είτε είναι πιο ακριβή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δίνεται επαρκής αιτιολόγηση. Υπάρχουν διάφορα σημεία σε λεπτομέρειε που θα μπορούσα να αναφερθώ, αλλά θα κοιτάξω να τα διατρέξω πιο γρήγορα. Για τι ε, υπηρεσίε Α και Β πάλι βλέπω εγώ κάποιε δυσκολίε. Νομίζω ότι μπορεί να περιπλέκει πολύ η κατάσταση και γι' αυτό θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι θα πρέπει να δούμε μέσα από τις διαπραγματεύσεις. Ξέρω ότι και χρονοβόρες είναι και κοπιαστικές καμιά φορά. Αλλά κύριε Ταραμπέλα, ας μην είναι μόνο η ιδεολογία αυτή που μας καθοδηγεί. Ας βρούμε και από την πρακτική ιδέες και λύσεις. Και ας επουστεύσουμε στο βαθμό που μπορούμε. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που μιλούν για απλοποίηση ε, πάση θυσία. Αλλά απλοποίηση η απλοποίηση που την υποστηρίζουμε έχει σημασία για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση πάνω απ' όλα. Αυτό θέλω να υπογραμμίσω. Το, μια περίπλοκη διαδικασία, μια περίπλοκη νομοθεσία μπορεί η μεγάλη επιχείρηση να την αντέξει και να την ακολουθήσει. Η μικρομεσαία όμως δεν είναι σε θέση να το πράξει πνίγεται μέσα στην ε, γραφειοκρατία και γι' αυτό πρέπει να απλουστεύσουμε τι ε, διαδικασίε έτσι ώστε να έχουν και μικρέ και μεσαίε επιχειρήσεις μια ευκαιρία επιβίωση. Ευχαριστώ κύριε Κρότσμαν. Η συντηρητική δεν εδώ, η CR, ο κύριος Διόγκ. Uh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή ο οποίος μελέτησε το θέμα με μεγάλη ταχύτητα. Συμφωνώ με τον ε, κύριο Σφάμπ που εκφράζει ανησυχίες. για κάποιες από τις αντιφάσεις, για τις κοινωνικές διαστάσεις, την ασφάλεια και το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίηση τους. Εγώ θα έχω περισσότερη δουλειά, διότι πρέπει να βεβαιωθώ και να βεβαιώσω ότι καθόλου δεν είχαμε αυτό το σκοπό. Είναι κρίμα. που οι δημόσιες σχέσεις μας δεν πέτυχαν το στόχο τους. Δώσαμε λαθασμένη εικόνα. Εδώ πρέπει να κάνω τις εξής παρατηρήσεις, ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε στις δημόσιες αρχές να εκπληρώνουν τις πολιτικές τους και να επιμένουν τις πολιτικές επιλογές που έχουν ε, αρχικά κάνει. Το είπε και η κυρία Ρούλε. Δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε στην νομοθεσία μας κατά λέξη τις δικαστικές αποφάσεις. Πολλές φορές υπήρξαν και πολλά επικριτικά σχόλια για, τις για συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις συγκεκριμένων υποθέσεων. Είναι λοιπόν ένα θέμα το θέμα της απλότητας και μετά υπάρχει και το θέμα των ανωτάτων ορίων. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα τα αυξήσουμε και κατά πόσον υπάρχει προστεθέμενη αξία για αυτό το είδους ε, τις νομοθετικές προτάσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και με περιφερειακές και τοπικές αρχές. Το σε τι κατάσταση έχουν περιέλθει και πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τα πράγματα και για εκείνους για το θέμα της απλότητας νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπαγορεύουμε στις ε, τοπικές και εθνικές αρχές πώς θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τον όγκο των ευθυνών τους και να μην ε, αναμειγνιόμαστε με τρόπο αντιπαραγωγικό. Επίσης ακούστηκαν και άλλες ανησυχίες που είχαν να κάνουν με την ε, δημοσιοποίηση. Θα πρέπει εδώ να είμαστε πολύ σαφείς. Συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Ρίλα για τους ορισμούς. Θα πρέπει να ορίσουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια τους στόχους αυτού του προγράμματος. Να δούμε τι ακριβώς επιδιώκουμε. Ποιοι είναι οι επιδιωκόμενοι στόχοι και όλα να οριστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλέσουν σάθα και προκύπτει μετά ένα σωρό δικαστικών διαφορών και υποθέσεων. Δεν θα επιμείνω τώρα σε σχόλια λεπτομεριών για τα επιμέρου κλάστερ, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξο και νομίζω θα καταλήξουμε σε συμβαστικέ λύσει παρόλο ότι μα περιμένει πολλή δουλειά. Ευχαριστώ. Α ακούσουμε τώρα άλλου βουλευτέ που ενδεχομένω θέλουν το λόγο. Τρει έχουν στήσει μέχρι τώρα, ο κ. Βαλτασάρε, ο κ. Ζιβό και ο κ. Βάιλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Ταραμπέλα για το τεράστιο έργο που έχει αναλάβει και για τους στόχους που έχει θέσει. Θα ήθελα να αντιληφθούμε ότι υπάρχει εξή συγκυρία, Ανδρέας. Δεν είναι οδηγία για τους δημόσιους διαγωνισμούς για τη Γερμανία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο αυτός. Όχι. Είναι μια οδηγία για 27 κράτη-μέλη. Καθένα από αυτά έχει τις δικές του αμφιβολίες, τα δικά του επικριτικά σχόλια, τα δικά του μειονεκτήματα και τις δικές του αρετές. Ποιος είναι λοιπόν ο στόχος που θέλουμε να πετύχουμε με την οδηγία αυτή. Είναι τελικός να προκοδοτήσουμε το ευρωπαϊκό σύστημα ε, δημόσιων διαγωνισμών με διαφάνεια που για λόγους λαϊκίστικους ή άλλους λόγους ε, δεν επιτυγχάνεται. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους ημετέρους ή αυτούς που δεν διαγωνίζονται με τρόπο ορθό. Θέλουμε να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Θέλουμε να ορίσουμε αρχές συστηματικότητας στους διαγωνισμούς. Νομίζω πως ναι. Θέλουμε οι δημόσιοι διαγωνισμοί να είναι ποιοτικοί, η διεξαγωγή τους να είναι ποιοτική. Θέλουμε να βραβεύσουμε και να, να τονώσουμε τις ε, υγιείς εταιρείε στην Ευρώπη. Με, που σέβονται τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, τα περιβαλλοντικά κριτήρια και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε σύγχυση στον όλο τομέα με όλα τα λάθη που μπορεί να διαπράξουμε και θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη του εγώ ίδιος το κάνω. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν είναι μόνο ιταλικό ελάττωμα το πρόβλημα στο κατασκευαστικό τομέα, είναι ένα πρόβλημα που είναι διαδεδομένο παντού. Άρα το κριτήριο της επιλογής μεταξύ εταιριών που σέβονται τις υποχρεώσεις τους και αυτές που δεν τη σέβονται, πέραν της ανταγωνιστικότητας, ακόμη και αν πρόκειται για περιπτώσεις του υποκόσμου, ξέρουμε πώς θα τις ε, αντιμετωπίσουμε. Ή θα τις λύσουμε ή όχι τις περιπτώσεις αυτές. Και αυτό στην Ιταλία, βέβαια, που εγώ γνωρίζω, αλλά θα μπορούσα να αναφέρω και τη Ρουμανία. Και φαντάζομαι ότι ανάλογε περιπτώσει μπορεί να προκύψουν και στη Γερμανία. Αυτή η διακριτική ευχέρεια που θέλουμε να συνεχίσουμε να διατηρούμε για τι δημόσιε αρχέ, με βάση ποιε εγγυήσει θα παράσχεται. Τη στιγμή που υπάρχει το ΕΜΗΡ με το άρθρο 169 για τις νέες προσφορές. Εάν μία εταιρεία κάνει προσφορά του 30% χαμηλότερη δεν πρέπει να τους ρωτήσουμε πώς σέβονται τις υποχρεώσεις τους. Τι σημαίνει όχι δεν θα βάλουμε όρια, δεν θα βάλουμε τίποτα και το αφήνουμε στη διακριτική ευχέρεια των δημοσίων αρχών. Ποιος θα μας αγγιηθεί ότι ο δημόσιος φορέας ε, εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι ένα συμφέρον μιας συγκεκριμένη επιχείρησης. Μα παρακαλώ δηλαδή, δεν είναι ότι θα ήθελα τα πάντα να τα καλύψουμε και να τα οχυρώσουμε, όμως αν θέλουμε διαφάνεια, ανταγωνιστικότητα, ισοτιμία, μπορούμε να το πετύχουμε. Το ίδιο και με το άρθρο 67. Με, το περιβό, με την περιβόητη αυτή διάτοξη. Η δική μου η μελέτη και οι δικές μου οι γνώσεις αφορούν και το δημόσιο δίκαιο, αλλά για τη χαμηλότερη τιμή αρκεί κανείς να έχει 15 ε, εργαζομένους που να τους κρύβεται να έρχονται ελεγκτές ε, εργασίας ή επίσης να παίζει με την ε, τιμή της βενζίνης και του πλαστικού αλλά τελικά δεν γίνεται έτσι η δουλειά Εάν λοιπόν αυτές τις τρευλώσεις δεν τις αντιμετωπίσουμε τι ακριβώς κάνουμε Ίσως να είναι υπέρμετρα τα και πολυάριθμα τα κοινωνικά κριτήρια. Όλα τα ραμπέλα είναι σοσιαλιστέ, αυτό να μην το ξεχνάμε. σω να είναι πρόβλημα τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Εντάξει, αλλά ο πυρήνα τη οδηγία είναι αυτό. Δηλαδή θέλουμε διαφάνεια και συστηματικότητα. Εντάξει για του ομίλου επιχειρήσεων, εντάξει για τι περιπτώσει υποδιαγωνισμών που τα πάντα ξοδεύονται. Και το λέω όχι γιατί είμαι υπέρ τη κρατική εξουσία, αλλά εντάξει πρέπει να υπάρχει και ελεκτική αρχή. Διότι αν μια γερμανική επιχείρηση θέλει να πάει στη Βουλγαρία για τι δραστηριότητέ τη, σίγουρα υπάρχει τάση να ευνοήσει κανεί τι ε, γειτονικέ περιπτώσει. Σε ποιον απευθύνεται αυτή η εταιρεία, εάν δεν έρθει αυτή η οδηγία να εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου απευθυνθεί η γερμανική εταιρεία σε δικαστήριο. Σε δικαστήριο γιατί δεν θα υπάρχει αρχή στην οποία να μπορεί να προσφύγει και να πει η οδηγία για τους δημόσιους διαγωνισμούς, η ενωσιακή οδηγία που ισχύει και στη Βουλγαρία και στην Ιταλία και στη Γερμανία προβλέπει το εξή. Και στην περίπτωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού ε, δεν έχουν καλυφθεί υποχρεώσεις. Θα επιληφθεί αρχή, δικαστική αρχή ή όχι. Θα πρέπει λοιπόν στις τοποθετήσεις μας, ε, τις αρχικές και μετά να προχωρήσουμε, χωρίς ιδεολογικά κολλήματα, να απαντήσουμε σε αυτές τις πτυχές, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει μία διάταξη και οικοδόμηση του, του νομοθετικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ιδάλλως δεν θα μπορέσει να γίνει, ιδίως λόγω της οικονομικής συγκυρίας που ζούμε. Ναι, κυρία Ρούλε, σας είδε. Αλλά φαντάζομαι ότι σε αυτό θέλετε κάποια παρατήρηση. Κύριε Ζουβά, αν επιτρέπετε να κάνει μια παρέμβαση, κυρία Ρούλε. Ναι, ήθελα απλώς να επισημάνω ότι έχουμε μια οδηγία για τα ένδικα μέσα και με αυτήν προβλέπεται επαρκής προστασία για τους διαδρομούς. Αν δεν λειτουργεί αυτή η οδηγία, αν τα δικαστήρια δεν λειτουργούν, τότε πρέπει να τροποποιηθούν τα δικαστήρια. Το ζήτημα δεν είναι όμω ζήτημα νομοθεσία, αλλά εφαρμογή σε εθνικό δίκαιο τη οδηγία για τα ένδικα μέσα. Πρώτον. Και δεύτερον, τα κριτήρια πρέπει να είναι ποσοστικά μετρήσιμα. Ποσοτικά μετρήσιμα, ώστε να μπορούν να τα επαληθεύουν τα δικαστήρια. Ιδάλω, πώ μπορεί το δικαστήριο να κρίνει Πρέπει να είναι σε θέση δηλαδή να δει νούμερα και να μπορέσει να κρίνει για να υπάρχει και η λογοδοσία και η επαλήθευση και ο έλεγχο. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Νομίζω ο κύριο Τουμπό ήταν εκείνο που είχε την οδηγία για τα ένδικα μέσα. Ομόφωνα την είχαμε κρίνει εδώ. Ήταν πολύ σημαντικό νομοθέτημα. Και τελικά δεν το γνωρίζει και κανένα. κύριο Σουβά έχει το λόγο. κύριε κυρία Πρόεδρε. Δύο-τρία ζητήματα θέλω να αναφέρω και πραγματικά συμπάσχω ε, με τον εισηγητή, γιατί εγώ είμαι από την άλλη πλευρά. Ξέρετε με ποιο θέμα ασχολούμαι. Πάρα πολύ καλά τα κατάφερε και στις εκλογές και τον συγχαίρω επίσης γι' αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων ε, επιχειρήσεων, ε, δεν είναι λεπτομέρεια το ζήτημα αυτό. Υπάρχει το περίφημο 90% της δραστηριότητας. Η έννοια δραστηριότητα είναι πολύ αόριστη. Τι θα πει δραστηριότητα. Είναι πόσα γεύματα σερβίρονται στη καντίνα, το κόστος των γευμάτων, ε, είναι πόσο πετρέλαιο καίει για να μεταφέρει το ψωμί από το αρτοποιείο στην κατίνα. Τέλος πάντων, ε, μήπως θα έπρεπε να λέμε 90% του κύκλου Αυτό είναι μια πρόταση που γίνεται στην οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης. Δεύτερο στοιχείο, στο άρθρο 11, πάλι για την ε, συνεργασία, φιλοσοφία μου είναι η ίδια. Νομίζω όμως ότι θα έπρεπε να προσθεθεί ένα νέο άρθρο που πολύ ξεκάθαρα και με σαφήνεια θα μιλά για την, τον, την εξαίρεση της μεταφοράς αρμοδιότητας μεταξύ τοπικών αρχών. Η γενική φιλοσοφία βέβαια αυτή είναι στο κείμενο, αλλά σήμερα όπως διαβάζουμε το κείμενο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Γι' αυτό και προσθέτω το 172 Euh, σε ό,τι αφορά την αμοιβαιότητα, τροπολογία ...1299 και 1302. Συμφωνώ με την αρχή της αμοιβαιότητας, αλλά αν δεν θέλουμε όλες οι δημόσιες συμβάσεις ε, να πηγαίνουν τα επόμενα 20 χρόνια σε Κινέζους, θα πρέπει να βρούμε νομικά στοιχεία που θα μας ε, δώσουν όπλα για να αμυνθούμε κι εμείς ε, αυτά τα οποία ε, βλέπονται στις τροπολογίες 1299 και 1302 είναι ένα είδος ε, ερζάτ σε έναν κανονισμό αμοιβαιότητας που μπορεί να μην και τόσο προφανής. Τρίτο σημείο. Ξέρω βέβαια ότι δεν είμαστε στο κλάστερ αυτό, σε αυτή τη δέσμη τροπολογιών, αλλά επειδή ετέθη το ζήτημα της εξαίρεσης των εταιριών υποψηφίων που έχουν καταδικαστεί για κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ε, αδικήματα. Τώρα, λέω, γιατί όχι, η ε, ίδια είναι η φιλοσοφία, απλά θέλω να είμαστε βέβαιοι ότι είναι τελεσίδικη η καταδίκη, ε, και όχι να έχει καταδικαστεί η εταιρεία μόνο και μόνο από ένα δημοσίευμα στον τύπο, γιατί κάποιε φορέ ε, τα μπερδεύουμε για αυτά τα πράγματα. Και υπάρχουν και οι εξή περιπτώσει. Παραδείγματο χάρη, μια εταιρεία στη Ρώμη καταδικάζεται για μια από τι θηγατρικέ τη, ή ένα τοπικό διευθυντή ε, πήρε κάποιε ελευθερίε με, τη... με το δικαίωμα συνεργασία και καταδικάστηκε η ίδια εταιρεία. Αντβίτα με τέρναμ πρέπει να αποκλείεται αυτή η εταιρεία από όλου του διαγωνισμού. είναι λίγο υπερβολικό σήμερα έχουμε για την IKEA, την πολύ μεγάλη εταιρεία αυτή, επειδή όλοι έχουμε επιπλατήσει στο σπίτι μας. Λοιπόν, στην Γαλλία υπάρχει ένα πρόβλημα με την εταιρεία IKEA. Ε, διώκεται στη Γαλλία η εταιρεία ε, γιατί ε, προβάλλει προσκόμματα στην αγορά εργασία. Τώρα δεν ξέρω αν καταδικάστηκε ή θα καταδικαστεί γιατί είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία. Επειδή όμω δύο-τρία άτομα στην διοίκηση τη εταιρείας στο Παρίσι είχαν μια πολύ προσωπική άποψη για τα δικαιώματα ε, τα εργασιακά θα πρέπει την οικία να την αποκλείσουμε από όλες τους διαγωνισμούς. Είναι πολύ πλοκό το ζήτημα αυτό. Και θεωρητικά συμφωνούμε, αλλά πρακτικά θα πρέπει να προσέξουμε να μην έρθει μπούμεραγκ. Να μην μπορεί δηλαδή να εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το οποίο θα προτείνουμε και αυτό θα είναι κρίμα και κακό και για το δημόσιο συμφέρον. Ευχαριστώ. So, äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορούμε να περιορίσουμε τη, τη, συζήτηση μάλλον χρονικά γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα αλλά από την άλλη έχουμε μέχρι τις 6.30 περιθώριο μόνο με την, ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως τον κύριο Ταραμπέλα, τον κύριο Σφάμπ ε, και θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε κάποια σημεία σημαντικά από τη μέχρι τώρα συζήτηση. Τα διαφιλονικούμενα κριτήρια που έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα, έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις, ότι είναι πλέον όριμη η εποχή για να οριστούν συγκεκριμένα πολιτικά κριτήρια, πράγμα που δεν είχε γίνει στο παρελθόν, γιατί δεν ήταν η ώρα του, δεν ήταν η εποχή του και δεν ήταν τόσο αποδεκτό. Εν τω μεταξύ όμω. πολλές εθνικές αρχές εισάγουν κριτήρια, έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου και από τον κύριο Μπαρνιέ ξέρουμε ότι και για την καινοτομία και για τα οικολογικά κριτήρια ε, θεωρούνται πάρα πολύ σημαντικά για τις συμβάσεις, λογικές συμβάσεις, τόσο για τη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες ξέρουμε ότι, θα πρέπει, ότι θεωρούνται πολύ σημαντικές και ότι πρέπει να γίνονται αποδεκτές ε, ως δεσμευτικές οι, οι συνθήκες τους, οι όροι τους. Αυτά τα κριτήρια. Τα άλλα κριτήρια, όσο πιο πολλά εισαχθούν, όπως πολύ συχνά όπως πολύ σωστά υπόθηκε, όσο πιο πολλά κριτήρια εισαχθούν, τόσο πιο αδιαφανής, ε, πιο αβέβαιη θα είναι η κατάσταση και πιο πολλά τα προβλήματα. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να το αφήσουμε σε μία σύσταση προς τις τοπικές αρχές, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, που θα πρέπει να αποφασίσει για ποιο συγκεκριμένο έργο, για ποια συγκεκριμένη σύμβαση, ποια κριτήρια θεωρεί πιο σημαντικά. Και έτσι, στην περιγραφή, στην προκήρυξη δηλαδή, μπορεί κανείς να γνωρίζει ότι οι ατάπετούμενα κριτήρια είναι αυτά. Για την ε, πιο φθηνή τιμή, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ πιθανό και άλλο λειτουργεί το σύστημα ε, να πει ε, μια δημοτική αρχή ότι προτιμεί, προτιμά όχι την πιο φθηνή προσφορά, αλλά αυτήν που παρουσιάζει τα πιο πολλά ειχέγγυα σε σεβασμού του περιβάλλοντος κτλ. Επομένως, πρέπει και αυτή η διάσταση να μην είναι ανοιχτή και να μην υποχρόνουμε για την ε, πιο φθηνή μόνο προσφορά. Για τον κύριο Μπαλτασάρε. Ιταλό συνάδελφο και όλους τους άλλους που ε, μίλησαν για την ε, Ιταλία. Όπως είπα, ήμουνα με την Επιτροπή Crime στην ε, Σικελία. Όλοι οι συνάδελφοι, οι Ιταλοί συνάδελφοι, αλλά και η Σικελία εκεί μας είπαν ότι δεν θα είναι εύκολο να ξεκινήσει μια διαδικασία για πιστοποίηση μη μαφιόζικων επιχειρήσεων ε, και βεβαίως δεν ε, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η μαφία έχει απλώσει τα πλοκάμια της σε όλες τις ε, χώρες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά, κύριε Ταραμπέλα, ίσως μια ιδέα θα ήταν να πούμε ότι εφόσον μια επιχείρηση έχει καταδικαστεί για εμπλοκή σε μαφιόζικες υποθέσεις, θα μπορούσε να αποκλειστεί από ένα διαγωνισμό. Αυτό όμως μπορεί να μου το απαντήσει την επόμενη εβδομάδα. Παρακαλώ τώρα η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους σκιώδης εισηγητές. Νομίζω ότι οι συναντήσεις πλέον των σκιωδών θα επικεντρωθούν στην ουσία. Απλώς γι' αυτό που λέγαμε για τους μισθούς και αυτό που έχει αποτελέσει ένα μεγάλο θέμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να ξαναδούμε τις διατάξεις για τις επιδόσεις των συμβάσεων, κάτι που στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποστηριχθεί ο ελάχιστος μισθός που δεν θα υπόκειται σε νομικούς περιορισμούς. Και δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί μια τοπική αρχή, μια εθνική αρχή, το ορίσιο ρήτρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση στον Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή για τον μισθό επιβίωσης όπως λέγεται, όχι τον ελάχιστο, τον μισθό επιβίωσης πολύ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ήθελαν αυτό να είναι πολιτικός στόχος. Είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι ο προηγούμενος Επίτροπος το 2009, απαντώντας στο κοινοβουλευτικό ερώτημα, είπε ότι είναι σημαντικό ο μισθός αυτός επιβίωσης να συνδυαστεί με, τις, ε, με τους δημόσιους διαγωνισμούς και τις ρήτρε επιχειρησιακής επίδοσης. Όμως, στις συναντήσεις των σκιωδών νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν ευρύτερα τα θέματα αυτά στο όλο πλαίσιο των διαδικασιών των δημόσιων προμηθειών. Κύριε Σβάμπ. Ναι, Πρόεδρε. Σε αυτή την παρατήρηση, κύριε Στάιλος. Θα ήθελα να, να απαντήσω στην κυρία Ρούιλα. Και να πω ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσει μια μεγάλη ποικιλία ε, όρων αμοιβή μισθών κτλ. Αλλά ή μη τι άλλο, ένα ελάχιστο όριο με βάση κάποιες λογικές συμβάσεις, όπως και αυτό το θέμα των ορφηγών που αναφέρατε εσείς, ε, ώστε να έχουμε ισότιμες συνθήκες εργασίας. Κύριε Αρούλε χωρίς μικρόφωνο. Καλώς, πολύ καλά. Συμφωνούμε λοιπόν, λέει ο κύριο Σφάπ. Θα δούμε πώς θα το διατυπώσουμε. Αυτό που θα μπορούσαμε επίση να κάνουμε θα ήταν να κάνουμε μια απευθείας παραπομπή στην οδηγία περί που ορίζει τις συνθήκες. Άρθρο 3, παράγραφος 8 για τον εργαζόμενο στην ε, οδηγία περί γιατί καλό θα ήταν να αποφύγουμε τις διαφορετικές ρυθμίσεις μεταξύ των δύο, δηλαδή τις ε, οδηγίες για τις συνάψεις των συμβάσεων και, αυτών, και αυτής περί αποσπάσεως. Ε, για δε την ε, κατηγοριοποίηση υπηρεσιών Α και Β, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει και η ομάδα μου προστίβεται θα πρέπει να τη διατηρήσουμε σε μια σειρά υπηρεσιών Μπορούμε ωστόσο, όπως προτείνει και ο κύριος Σταραμπέλα και άλλοι συνάδελφοι, να διατηρήσουμε ένα βαθμό ευελιξίας τα επιχειρήματα για τις υπηρεσίες είναι σημαντικά. Υπάρχουν ε, κράτη όπως η Ιταλία, νομίζω, κύριε συνάδελφε, για τα οποία η υπηρεσία πολιτικής προστασίας έχει μάλλον ε, στρατιωτική δομή, ενώ άλλες έχουν πιο πολιτική δομή. Πες μια λίστα πρέπει να βρεθεί. Για τον κύριο Παλτασάρ επίσης ε, επισήμανε ότι οι διατάξεις που θα εισαχθούν θα ισχύουν για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι για ένα κράτος μόνο. Και αντίστοιχα θα πρέπει να είμαστε σε θέση και να παρακολουθούμε την εξέλιξη της νομολογίας. Δηλαδή χρειάζεται μια ε, ενημέρωση, μια ροή ενημέρωσης, μη γραφειοκρατική, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, όταν μιλούμε για προσφορές, θα πρέπει να, να κρίνονται αυτές όχι μόνο με βάση το κόστος, αλλά να επιλέγονται πάντα οι καλύτερες προσφορές. Κύριε Πρόεδρε, και αυτό είναι το τελευταίο σχόλιο. Έχουμε προχωρήσει, πιστεύω, αρκετά. Είμαστε πολύ κοντά στην ψηφοφορία. Ίσως είναι δύσκολο να ε, δώσουμε νέες διατυπώσεις για όλες τις πιθανές τροπολογίες. Ελπίζω πάντως ότι ο κύριος Ταραμπέλα και οι σκιώδεις συγκητές θα μπορέσουν να εργαστούν εντατικά ώστε να βρούμε στο δυνατόν πιο αρμονική και αποδεκτή λύση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Πάολα Τζανέτη. Ευχαριστώ. Τρία σε μία πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα για τις υπηρεσίες. Να επιβεβαιώσουμε εδώ μια βασική αρχή που καμιά φορά χάνεται στη συνέχεια της συζήτηση από το α προς το β και για τις υπηρεσίες, για την οδηγία αυτή και την, ε, αυτή που έχετε μπροστά σας και την μελλοντική της εκδοχή. Οι υπηρεσίες δεν καλύπτονται από την οδηγία ανακατηγορία δεν υπάρχουν ήδη υπηρεσιών που καλύπτονται και άλλα που δεν καλύπτονται. Δεν μας ενδιαφέρουν τα είδη των αγορών, αλλά ο τρόπος που είναι διοργανωμένε. Δηλαδή, τι... μας ενδιαφέρουν οι συμβάσει που διέπουν τι υπηρεσίες. Εάν είναι ιδιωτικέ δημόσιες, εάν ε, έχουν ε, ανατεθεί σε εξωτερικό οικονομικό συνεργάτη βάσει διαγωνισμού, εάν υπάρχει αμοιβή ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση εμπίπτουν στην οδηγία οι υπηρεσίες αυτές. Θα μπορούσε να είναι και είδους α και τύπου α και τύπου β ή βάσει της οδηγίας οποιαδήποτε υπηρεσία, ιδίως στο παράρτημα 16, κοινωνικές υπηρεσίες, υγειονομικές και ούτω καθεξής. Όμως όλες μπορούν να έχουν σχέση με την οδηγία, εάν έχουν ε, ανατεθεί βάση δημόσιου διαγωνισμού. Εάν έχουν να τεθεί βάση νόμου ή με άλλο τρόπο ή υπάρχει in-house διοργάνωση και η αναθέτουσα αρχή η ίδια το έχει καθορίσει, δεν εμπίπτουν στην οδηγία σε όποιο τύπο και να ανήκουν. Άσχετα με το τι λέει το παράρτημα 16 για τα είδη ή όχι. Να το ξεκαθαρίσω αυτό επίση εξ αρχή, γιατί καμιά φορά το ξεχνάμε όταν συζητάμε για τι κατηγορίε Α και Β. Όλε λοιπόν οι υπηρεσίε θεωρητικά μπορούν να καλύπτονται την οδηγία και αυτό που καθορίζει το αν εμπίπτουν ή όχι είναι ε, ο τρόπο που έχουν ανατεθεί. Τώρα, η κατηγορία του, το παράρτημα 16 και κατά πόσον ισχύουν όλα αυτά έχουν σημασία μόνο για το σύστημα που εφαρμόζεται για την ε, ανάθεση. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή για να φτάσουμε στον ορισμό των καλύτερων δυνατών κανόνων. Είναι σημαντικό όμως οι κανόνες αυτοί να εφαρμόζονται. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι οι κανόνες δεν εφαρμόζονται αρκετά σωστά. Το επίπεδο πλημελούς εφαρμογής το επίπεδο σφαλμάτων είναι πολύ ψηλό και για τερθωτικούς λόγους. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολλές διατάξεις που αφορούν τη διακυβέρνηση. Τώρα οι δομές, τα όργανα, η διοργάνωση είναι σαφές ότι μπορούν να το καθαρίσουν, να το καθορίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κάτι μέλη. Θα διαχειριστούν το όλο θέμα μόνοι τους, αλλά θα πρέπει να οριστεί ένας κατάλογος υποχρεώσεων. Κάποιες επαληθεύσεις που θα πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστούν η απάτη, η διαφθορά και ούτω καθεξής και για να υπάρχει ορθή εφαρμογή των κανόνων. Τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι κάτι που αφορά το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα μόλις περιμένουμε το τέλος ε, της ομάδας εργασίας, συζητήσεων στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για το θέμα των δημόσιων προμηθειών και θα εξεταστεί το κείμενο της κλασικής οδηγίας, το ενοποιημένο κείμενο και την επόμενη εβδομάδα θα γίνει συνάντηση για να συζητηθεί η οδηγία για τους ηθικούς τομείς και αυτά εν ώψη του Κορεπέρ στις 21 Νοεμβρίου. Εκεί κατά πάσα πιθανότητα θα ανατεθεί εντολή τουλάχιστον για την κλασική οδηγία. Αυτά ενημερωτικά. Και τέλος, οι υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι στη διάθεσή σας για τεχνικές διευκρινήσεις, για τις συζητήσεις που θέλετε να κάνουμε και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μαρκ για να κλείσει. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, για να τα πάρω με τη σειρά. Πρώτη παρέμβαση, ΣΦΑΠ. Υπήρξε μια δήλωση στον τύπο. Μην εστιάζετε όμως τόσο πολύ σε αυτή τη δήλωση, γιατί δεν ήταν γενική, αφορούσε πολύ συγκεκριμένα μια λεπτομέρεια που έχει τη σημασία της παρόλα αυτά, γιατί γνωρίζουμε συχνά ότι παλιά, δεν θέλω βέβαια να κατηγορήσω την Επιτροπή και γνωρίζω ότι ο Επίτροπος Μπαρνιέ θέλει τις ε, δημόσιες αρχές να τις διατηρήσει σε ένα ύψος, να έχουν τις δυνατότητες που πρέπει να έχουν και σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θέλω να πω τίποτα, αλλά έχει και κάποιου υπαλλήλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια δεν ε, αναφέρουμε στην κυρία Ζανέτη. Αλλά ξέρετε, μπορεί οι επίτροποι να φεύγουν, αλλά παραμένουν υπάλληλοι. Μεταξύ αυτών είναι κάποιοι εξαιρετικοί, αλλά κάποιοι παρά τη επικαιρότητα, παρά ε, την πραγματικότητα, θέλω να τα ιδιωτικοποιήσουν όλα. και μπορεί ε, αυτοί να εργάζονται για δεκαετίες ακόμη. Αυτό που δεν συμφωνώ και ήθελα να αφισβητήσω είναι κάτι που ίσως να ίσχυε στις προηγούμενες οδηγίες. Δηλαδή, στο άρθρο 74 του σχεδίου οδηγίας λέγεται ότι τα κράτη-μέλη, όσο τα επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν σε διαγωνισμό όλες τις υπηρεσίες που υπάγονται στο παράρτημα 16. Διαβάζοντα το παράρτημα 16, αυτό μπορεί να φανεί λεπτομέρεια, γιατί μιλάμε για παράρτημα, αλλά υπάρχει ένα εδάφιο που λέει κοινωνική ασφάλιση, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση των κρατών μελών. Εκεί λοιπόν πράγματι αντέδρασα, πραγματικά ενοχλήθηκα, γιατί δεν θα ήθελα ε, αφού θέλουμε να βελτιώσουμε την οδηγία για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, να μπορεί κανείς να κατηγορήσει εμάς και εμένα προσωπικά ως εισηγητή ότι σε ένα εδάφιο προβλέπω ήδη τη μελλοντική ιδιωτικοποίηση τη πολιτική κοινωνική ασφάλεια των κρατών μελών. Όταν λοιπόν κάποιο εδώ μου προσάπτει ότι θέλω να νομοθετήσω, βελτιώσω την οδηγία για να προσπαθήσω να βελτιώσω τις διαδικασίες και να αποφύγω την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με όχι στο σωστό τρόπο, που σήμερα μέσω του dumping όταν έχουμε δηλαδή διαδοχή των ε, αναδόχων που δεν είναι με τρόπο διάφανο. Μου λένε λοιπόν και μου προσάπτουν ότι θέλω να παρέμβω στι κοινωνικέ πτυχέ και τα κοινωνικά συστήματα. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ, όχι μόνο προ ε, το συμφέρον των εργαζομένων, ως μέλος των σοσιαλιστών μπορεί κανείς να μου πει ότι είμαι πιο ευαίσθητος σε ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αλλά εγώ μιλάω και για τους ε, εργοδότες και τις επιχειρήσεις που σήμερα πλήττονται από αθέμπτο ανταγωνισμό, ιδίως στον τομέα της οικοδομής, των υπηρεσιών καθαριότητας, ε, των μεταφορών που... Ε, και έχουμε και την ε, διαδικασία της απόσπασης των εργαζομένων που προσλαμβάνουν εργαζομένους ε, ε, χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα που εργάζονται με μαύρη εργασία. Αυτή ε, πρέπει να του προστατεύσουν και θα πρέπει να έχουμε ένα εργαλείο που θα μας επιτρέπει να έχουμε την εξυγίανση των δημοσίων συμβάσεων αλλά με την εμβόλια και κυρώσεων. Και θα πάνω σε κάτι που είπε ο Φιλίπ Ζιβά. Απέναντι λοιπόν στι επιχειρήσεις που δεσάβονται του τους κανόνες του παιχνιδιού. Και πρέπει να έχουμε κοινωνικά κριτήρια και να σεβόμαστε τα, τα, τους όρους του παιχνιδιού. Έχουμε την Σύμβαση 94 ε, της Διεθνούς Οργάνωσης, Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που δυστυχώς δεν την έχουν ε, επικυρώσει παρά 11 κράτη-μέλη. Τουλάχιστον να την εφαρμόσουν αυτοί που την έχουν επικυρώσει, αλλά και τι οδηγίε και το εθνικό δίκαιο και τι ε, συλλογικέ συμβάσει εργασία που έχουν ισχύ νόμου και αν υπάρχει και συμφωνία μεταξύ εργοδότη και συνδικάτου και αυτό πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να αποφύγουμε το κοινωνικό dumping πήρα μια πολύ ενδιαφέρουσα εξήγηση από τον Επιτρόπο στο Στρασβούργο για το άρθρο αυτό. Αυτό που ζητώ εγώ είναι διευκρινήσεις απλά από την Κομισιόν για το άρθρο, για το παράρτημα 16 που αναφέρεται στο άρθρο 74 και όπως είπατε κύριε ΣΦΑΠ και στο άρθρο 10 υπάρχει τροπολογία που λέει εξαίρεση της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης από το πεδίο εφαρμογή οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις. Τώρα, έρχομαι σε άλλα σημεία τα οποία αναφέρατε. Για τη διακυβέρνηση μπορώ να πω ότι χονδρικά εξαιρουμένου ενός σημείου, νομίζω ότι προχωρούμε καλά. Θα μιλήσω ε, πιο αναλυτικά για τους κοινούς ορισμούς όταν αναφερθώ στα σχόλια του κυρίου Ζιβά πράγματι για τις διοδηγίε, είτε είναι τομεακέ είτε είναι γενικέ, για τις συμβάσει σε παραχώρηση και για τις δημόσιε συμβάσει πρέπει να τα δούμε. Εγώ είμαι εισηγητής για τις δημόσιε συμβάσεις βέβαια. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το, τις συλλογικές συμβάσεις. Η αναφορά στι συλλογικέ συμβάσει ε, που γίνεται από το ΕΛΚ είναι θετική ε, αλλά αναφέρεται μόνο στι συλλογικέ συμβάσει που δηλώνονται και ισχύουν καθολικά. Όμως η, οδηγία, η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων που αναφέρατε και εσείς και το ΕΛΚ Μιλάω για τι γενικά εφαρμοστές συλλογικέ συμβάσει, αλλά και αυτές που συνάπτονται μεταξύ κοινωνικών εταίρων, των πλέον αντιπροσωπευτικών κοινωνικών εταίρων, όπως λέει. Για τη δική μας ομάδα, όλες οι κατηγορίες πρέπει να καλύπτονται και πρέπει να γίνονται σεβαστά ε, τα ενωσιακά δικαιώματα και οι πρακτικές στα κράτη-μέλη. Ο κ. Μπαλτασάρη είπε ότι δεν κάνουμε μια οδηγία για τη Γερμανία, τη Σουηδία, το Λουξεμβούργο, αλλά θέλουμε να είναι εφαρμόσιμη σε όλα τα κράτη-μέλη και θέλουμε να υπάρξει μια σύγκληση των κανόνων για την κυρία Ρούλε. Δεν κατάλαβα πολύ καλά τι είπε η κυρία Ρούλε. Λέει ότι αναθέτουσα αρχή πρέπει να έχει ασφάλεια. Συμφωνούμε να υπάρχουν κάποιε διασφαλίσεις. Και είπατε ότι έχετε επαφέ με τι τοπικές αρχές και ότι σας είπαν ότι η φθηνότερη προσφορά είναι, καλή, ε, είναι το καλύτερο για την ασφάλεια. Εάν περιοριστούμε σε αυτό, ε, δεν συμφωνώ. Δεν ξέρω αν ε, συμφωνεί μαζί σας και, και η υπόλοιπη ομάδα σας. Θα μιλήσω με τους συναδέλφους σας πάντως, αλλά Εμεί είμαστε κατά τη δικτατορία χαμηλότερη χαμηλότερης τίμης προσφοράς που παραγνωρίζει δικαιώματα σε ό,τι αφορά κοινωνικά δικαιώματα, περιβαλλοντικά αισθήματα κτλ. Όπω είπατε θα πρέπει να επικεντρωθούμε στι υπηρεσίε που έχουν τοπικό χαρακτήρα, αλλά και εγώ μίλησα με την νορβηγική κυβέρνηση και συμφωνούν μαζί μου. Με την αναφορά δηλαδή ε, στη Σύμβαση 94 της Διεθνής Οργάνωση εργασία. Οργάνωσης Εργασίας. Είναι μια χώρα που προστατεύονται τα κοινωνικά δικαιώματα και που μπορεί να πέσουν θύματα εκεί ε, του κοινωνικού ντάμπινγκ. Γι' αυτό με οι Νορβηγία. Του συνάντησα, ίσως ήταν ε, λίγο πριν από εσά ή λίγο μετά από εσά πάντως χαίρονταν πάρα πολύ με τι απόψεις μου. Τώρα για τον κύριο Κρότσμαν ε, έχετε κάποια αμφιβολία. Α, δεν είναι εδώ ο κύριο Κρότσμαν, είναι εδώ, είναι. Λοιπόν, σα περιμένω για να βάλετε τα ακουστικά σα να ακούσετε τη μετάφραση. Λοιπόν, έλεγα κύριε Κρότσμαν, ότι η αμφιβολία που εκφράστηκε για την απλούστευση με βρίσκει σύμφωνο, δεν θα τα καταφέρουμε, είναι σαφέ. Θέλουμε να απλουστεύουμε συνεχώ και δεν το καταφέρνουμε. Κρίμα είναι αυτό, αλλά. Όταν πρότεινα έτσι κάπω ε, ριζοσπαστικά, φυσικά και πρέπει να έχουμε καινοτομία, πρέπει να, δώσουμε, να βρούμε χώρο για την καινοτομία, αλλά και για την εταιρική σχέση, για την καινοτομία, για τον για ανταγωνισμό φυσικά. Αλλά όταν μιλάμε για ανταγωνιστικό ε, διάλογο, πώ θα το εφαρμόσουμε χαιρετίσματα. Θα είναι δύσκολο, διότι σε κάποια ε, τομείς λειτουργεί, σε κάποιους όχι. Και πρέπει να έχουμε τα, τα, τα, τα λόγια να τα κάνουμε έργα, αλλά τουλάχιστον πρέπει να τα βάλουμε στο χαρτί. Δεν ξέρω αν είναι μια χαμένη μάχη από την αρχή. Είναι πάντως αυτά, τα λέμε στην έκθεση και υπάρχει χώρος και για την καινοτομία και για τον ανταγωνιστικό διάλογο, για να υπάρχει καλύτερος και γέστερος ανταγωνισμός. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απλούσευση των διαδικασιών για τις ΜΜΕ, μεγάλη, είναι με ένα μεγάλο μέλημα για μένα και για τις αναθέτουσες αρχές κυρίως. Αυτές πρέπει να χωνέψουν, αν θέλετε, και να εφαρμόσουν την οδηγία. Αν δεν απλουστεύσουμε και την ίδια τη ζωή των αναθετουσών αρχών, θα έχουμε χάσει τον βασικό στόχο. Και βέβαια χρειάζεται απλούστευση και για τις επιχειρήσεις. Νομίζω είναι η δέσμη 4 που μιλάει για, για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ή procurement. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να είναι δεσμευτικέ οι διατάξει, Γιατί θέλουμε να υπάρχει απλούστευση, αλλά και μικρομεσαίε επιχειρήσει να μπορούν να συμμετέχουν και πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα σε μια σειρά δημοσίων συμβάσεων να ενημερώνονται με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα για δυνατότητε που τους διαφεύγουν. Είναι λοιπόν μια πύλη εισόδου για την καλύτερη συμμετοχή των ΜΜΕ ε, στους δημόσιους διαγωνισμούς. Για τον κύριο Ντε που εξέφρασε και αυτό στην ανησυχία του για τις κοινωνικέ υπηρεσίες, τον κίνδυνο να ιδιωτικοποιηθούν κτλ. Θα προσπαθήσουμε να το περιορίσουμε τον κίνδυνο αυτό, αλλά υπάρχει μια τάση σήμερα γενική που δίνει τη δυνατότητα ε, στις δημόσιες αρχές να μπορούν να οργανωθούν και ο Φιλίπ Σιβά συμβάλλει σε αυτό, στο να μπορεί να γίνει αυτό με κάποιου όρου και προποθέσει, αλλά να έχουν οι δημόσιε αρχέ πάντω και κάποια αυτονομία και να μπορούν να οργανώνουν τι υπηρεσίε του όπω ε, κρίνουν σκόπιμο. Να πρέπει να συνεχίσουν να φέρουν σε πέρα στην αποστολή του αναθέτου τη αρχέ. Φυσικά και συμφωνώ. Αναφερθήκατε επίση και εσεί στην απλούστευση. Σίγουρα είναι δύσκολο το να προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε. Δεν θέλω βέβαια να κατηγορήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να απαντήσει η κυρία Ζανίτη βέβαια, αλλά ω εισηγητή και με του σκιώδει είχα το πλεονέκτημα ότι εξεργάστηκα ένα σχέδιο οδηγία που συνολικά είναι καλό, πηγαίνει προ την καλή κατεύθυνση και δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό στο Κοινοβούλιο. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να διορθώσει και πολλά πράγματα γιατί είναι καλή πορεία. Μπορούμε να συμφωνήσουμε επί τη ουσία στα πιο σημαντικά αλλά εκτιμούμε διαφορετικά κάποιες πτυχέ. Αυτό πρέπει να είναι γνωστό για τον κύριο Μπαλτασάρε που έπρεπε από αυτό να ξεκινήσω και να τον συγχαρώ. Να συγχαρώ και την πρόεδρο που δεν τον διέκοψε τον κύριο Μπαλτασάρε παρότι μίλησε για αρκετή ώρα. Και να ε, συμπεριλάβω και την κυρία Πίτη Θα είναι εύκολο, πιστεύω, με τις δικές σας ε, προτάσεις να ε, καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση. Ο βασικός στόχος μας εδώ είναι η ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων να γίνει πιο σωστά. Οι αναθέτουσες αρχές ε, που θέλουμε να διευκολύνουμε είναι ουσιαστικά εκπρόσωποι των πολιτών που θέλουν να θέσουν δημόσιες συμβάσεις για υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και με χρήση δημοσίων κονδυλίων που θα πρέπει να είναι το πλέον αποδοτική δυνατή. Αυτό είναι ο βασικό στόχο αλλά βέβαια πρέπει να ωφελείται και η πραγματική οικονομία. Επιχειρήσει να μπορούν να υποβάλουν τι προσφορέ του με σαφή διαφανή τρόπο χωρί να υπάρξει διασπάθηση χρημάτων. Κυρία Βάιλερ μίλησε για τη μαφία. Και είπατε ότι δεν υπάρχει σε όλε τι χώρε. Μα όχι, υπάρχει. Παντού είναι παρούσα. σω να είναι λιγότερο ορατή η παρουσία τη σε κάποιε χώρε, αλλά η μαφία, οι μαφίε, οι κλιματικέ οργανώσει υπάρχουν και είναι παντού. Δεν περιορίζονται στη και για, για να μιλήσω για πολιτική για τη δευτερόλεπτα, εκλέχθηκε ένας περιφερειάρχης που δεν έχει σαφή πλειοψηφία και θα έχει δύσκολο έργο, αλλά είναι κάποιο που ε, συμβολίζει την μάχη κατά της μαφίας. Ο Ζάρη Γκροσέτα είναι ο συναδελφός μας, ε, το ξέρουμε τι έχει περάσει και τι περνάει. Λοιπόν, παράθεση ήταν αυτή. Κύριε Ζιβά, συνεργασία δημόσιων επιχειρήσεων. Δεν ήταν σαφή, έτσι όπως τα είπα και για τα ποσοστά, πράγματι θα τα διευκρινίσω, για να μπορεί να μου προσάψει κανείς τίποτα. Σε ό,τι αφορά την αμοιβαιότητα. Και αυτό μπορεί να συζητείται αλλού, ναι, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Πρέπει να εγγυηθούμε την αμοιβαιότητα, γιατί γενικά, και το δείχνουν και τα στοιχεία, όλοι οι οικονομικοί παράγοντες σημαντικότεροι είτε σε βιομηχανισμένες είτε σε αναδυόμενες χώρες εδώ και καιρό είναι υπέρ του ανοίγματο. Καλό αυτό. Άλλοι όμω εφαρμόζουν, άλλοι δεν εφαρμόζουν το άνοιγμα αυτό. Και χρειάζονται τα εργαλεία τη αμοιβαιότητα. συμφωνώ. Έτσι, οι σχέσει μεταξύ των διαφόρων μπλοκ ε, σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι ισορροπημένε. και δεν θα έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό. Άλλοι δηλαδή να μπαίνουν στι δικέ μα αγορέ και εμεί να μην μπορούμε να τι στις δικές Θα Συμφωνώ πολύ σωστά. Είπε ότι αν κάποιος, μια επιχείρηση στη Ρώμη καταδικαστεί για μια παραβίαση ενό εργασιακού δικαιώματο, θα πρέπει αυτό να συνεπάγεται τον αποκλεισμό τη διαβίου από όλε τι ε, συμβάσει. Δεν μπορεί ένα υπάλληλο ή ε, κάποιο να θέτει σε κίνδυνο την εταιρεία και να μην τη επιτρέπει να συμμετέχει σε διαγωνισμού. Είτε στη χώρα της είτε σε άλλες χώρες. Ο Φρανκ Έγγελ βρήκε μια ενδιαφέρουσα διατύπωση, το είπε και για την Μπάρμπαρα Βάιλερ, νομίζω στην τελευταία τη ερώτηση, αναφέρθηκε σε μια εταιρεία ε, η επιχείρηση η οποία αναγνωρίζεται ως ένοχη και πώς ορίζουμε αυτό. Μιλάμε για σοβαρό αδίκημα και επαναλαμβανόμενο αδίκημα. Σοβαρό και επαναλαμβανόμενο. Αυτό για να αποφύγουμε μία υπόθεση με απόφαση ενός ε, δικαστή σε μία χώρα να εξαιρεί, να αποκλεί την επιχείρηση από τη συμμετοχή της σε συμβάσεις. Είναι ενδιαφέρουσα λοιπόν αυτή είναι. Τώρα η κυρία Βάιλερ μίλησε για τα κριτήρια. Είπατε ότι είναι ε, όριμη στιγμή για να ε, μιλήσουμε για στρατηγικά κριτήρια, περιβάλλον, συλλογικές συμβάσεις κτλ. Είπατε όμως ότι θα πρέπει να αποφασίζει ο Δήμαρχος και το επιτέλειο. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Γερμανία, αλλά στο Βέλγιο μόνο ε, ένα μικρό μερίδιο εξουσίας έχει ο Δήμαρχος. Ουσιαστικά ε, όλοι μαζί. Το Κοινοτικό Συμβούλιο ορίζει τις ε, προϋποθέσεις του όρους των διαγωνισμών, στο Βέλγιο παραλαμβάνω, και στη συνέχεια όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ε, θα χειριστεί τη διαδικασία. Διαβούλευση, ανάθεση, κατακύρωση της σύμβασης, όχι μόνο στο Δήμαρχος, για την κυρία Στάιλερ, για τον κατώτατο μισθό όπου υπάρχει. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνονται σεβαστέ οι συλλογικέ συμβάσει εργασία και οι νόμοι όπου υπάρχουν. Είναι σημαντικό αυτό. Και για να ολοκληρώσω, επανέρχομαι στον κύριο Σφαπ και στην κυρία Ζανέτη. Αρμονική ψηφοφορία. Ναι, θα μπορούσε να το πετύχουμε. Είχαμε διάφορες συναντήσεις. Ε, έχουμε αυτούς τους συμβιβασμούς που δεν είναι όμως ε, ακόμη εξασφαλισμένοι. Α, δεν θέλετε να πείτε αυτό. Α, ναι, γιατί ε, είχαμε πράγματι πρόοδο μετά από τις πολλές συναντήσεις με τους Κιώδης. Κάναμε βήματα προς κατεμέ αποδεκτούς συμβιβασμούς και όχι μόνο κατεμέ, φαντάζομαι, γιατί συμφωνήθηκαν οι συμβιβασμοί από τις διάφορους και περισσότερου περισσότερους τουλάχιστον από αυτούς. Άρα εγώ δεν απελπίζομαι προσωπικά. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα που ανέφερε η κυρία Ζανέτ στην παρέμβασή τη, εγώ χαίρομαι που στο Συμβούλιο που ούτε και εκεί ήταν εύκολα τα πράγματα, γιατί θυμάμαι όταν αναφερθήκαμε για πρώτη φορά στο χρονοδιάγραμμα ΙΜΚΟ και μιλήσαμε για ψηφοφορία στι 10 Οκτωβρίου, αυτό ήταν το πρώτο χρονοδιάγραμμα στην Επιτροπή μα, λαμβάνοντα υπόψη όλε τι προθεσμίε, κατάσταση τροπολογιών τον Ιούλιο, μετάφραση, 2.500 τροπολογίε να μεταφραστούν, μετά να τι επεξεργαστούμε σε ομάδε εργασία ε, και στην Επιτροπή μα αλλά και σε επίπεδο σκιωδών. Μην ξεχνάμε και τις 7 επιτροπές που γνωμοδοτούν, που έχουν ή θα γνωμοδοτήσουν. Ήταν λίγο δύσκολο να τηρήσουμε λοιπόν αυτό, αυτή την προθεσμία της 10 Οκτωβρίου. Μας λέγαν όμως ε, στην Κομισιόν ότι μάλλον το μάθα θα φτάσει στο Συμβούλιο σε εκείνη γνώμη και ξέραμε ότι δεν είναι σε εκείνη θέση γνώμη. Αυτό το ξέραμε ότι ήταν δύσκολο και αποδείχθηκε αδύνατο σήμερα. Δεν ξέρω αν ε, ε, στην 21η Νοεμβρίου θα υπάρξει συμφωνία σε επίπεδο κορυφαίρα σε επίπεδο Συμβουλίου. Εμείς είπαμε 28-29 Νοεμβρίου για την κλασική οδηγία στην Επιτροπή μας και 18 Δεκεμβρίου ΜΕΑΚΙ. Πέντε μήνες προβλεπόταν αρχικά να είναι διαφορά, από το Μάιο για το Συμβούλιο και τον Οκτώβριο για την ΙΜΚΟ, φτάνουμε τελικά σχεδόν ε, ταυτόχρονα να αποφασίζουμε. Και αυτό θέλουμε. Θέλουμε η οδηγία ε, να μπει κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τουλάχιστον στο κοινοβούλιο. Να έχουμε αυτό το δωράκι για τις γιορτές και μετά έχουμε και τους τριμερείς διαλόγους που με βέβαιος ότι θα είναι αρκετά φορτισμένοι και ζωντανοί. Αυτά είχα να πω σε αυτή τη φάση κυρία Πρόεδρε απαντώντας στους διαφόρους συναντέλους. Ευχαριστώ. vielen Ευχαριστώ κύριε Ταραβέλα. διεξοδικά απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Έχουμε διευκρινίσει νομίζω ότι ήταν εκκρεμές. Και εύχομαι καλή συνεργασία μέχρι τις 29 Νοεμβρίου με τους συναδέλφους σας για να γυρίσουμε μετά στην Επιτροπή για την Ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ και αύριο το πρωί τα ξαναλέμε.